Bene. Cominciamo. Ας αρχίσουμε. Καλημέρα σας. Έχουμε πολλές συναντήσεις σήμερα. Άρα δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε παρόλο που λείπουν αρκετοί συνάδελφοι. Πρώτο, το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορά την έγκρισή της. που έχετε στους φακέλους σας. Εάν δεν υπάρχουν επιφυλάξεις ή παρατηρήσεις, εγκρίνεται η μερίσια διάταξη χωρίς αλλαγές. Σημείο 3. Έγκριση των πρακτικών. Έχετε τρία πρακτικά στους φακέλους σας. Εάν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, θεωρούμε ότι τα πρακτικά εγκρίνονται. Περνάμε στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την ενεργειακή απόδοση του εξοπλισμού γραφείου που τροποποιεί έναν κανονισμό. και την συμφωνία μεταξύ ΙΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον συντονισμό προγραμμάτων ενεργειακής απόδοσης. Δίνω το λόγο στην κυρία Μπέλα Κόβατς, στην εισηγήτρια. Τον κύριο, με συγχωρείτε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένε Πολιτείε το 2000 υπέγραψαν μια συμφωνία για το συντονισμό των, ε, της τυποποίησης του εξοπλισμού γραφείων, ο οποίος παρατάθηκε το 2006 για άλλα πέντε χρόνια. Θέλει λοιπόν να εισαχθεί το Energy Star Program στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή η συμφωνία. Το προβλέπει. Μαζί λοιπόν με την υπηρεσία για το περιβάλλον της, ε, ε, των Ηνωμένων Πολιτειών και τις δικές μας υπηρεσίες προσπαθούμε να καθορίσουμε προδιαγραφές για προϊόντα και τα εγκεκριμένα προϊόντα να χρησιμοποιούνται μετά ε, και στις δύο πλευρές και να αναγνωρίζονται αμοιβαία. Το πρόγραμμα αυτό πέρασε το 2008 μέσω του κανονισμού 106. Το πρόγραμμα αυτό συνέβαλε ούτως ώστε η αγορά για τον εξοπλισμό των γραφείων να λαμβάνει περισσότερο υπόψη την ενεργειακή αποδοτικότητα και επίσης υπήρξαν εξοικονομήσεις για τους καταναλωτές μεταξύ 2008 και 2011 το πρόγραμμα Energy Star είχε ως αποτέλεσμα να μειώσουμε κατά 16% την ενεργειακή κατανάλωση στα γραφεία και σύμφωνα με εκτιμήσεις το πρόγραμμα αυτό μέχρι το 2020, θα μειώσει την κατανάλωση ενέργειας στα γραφεία ε, γύρω στο 30%. Πριν λοιπόν λήξει το πρόγραμμα το Δεκέμβριο του 2011, ξεκίνησε η Κομισιόν διαπραγματεύσει με τι ΗΠΑ, ούτω ώστε να καταλήξουν σε νέα συμφωνία και να επιμηκύνουμε το πρόγραμμα για πέντε χρόνια και μέχρι τέλους του 2011 έκλεισαν αυτές οι διαπραγματεύσεις. Πρώτα απ' όλα λοιπόν πρόκειται για τεχνικές προσαρμογές. Οι αλλαγές δηλαδή αφορούν τεχνικές προσαρμογές, οι προτινόμενες τροπολογίες. Για παράδειγμα, ε, ενημερώνονται οι παραπομπές στο, στο ισχύον δίκαιο, οι περιεχόμενες αλλαγές είναι ότι θα υπάρχουν δύο διαφορετικά συστήματα ε, ε, τυπο, ε, χορήγησης ε, αδειών. Έγκριση δηλαδή. Εμείς ε, στην Ευρώπη προτιμούμε να εγκρίνουμε να, τη διαδικασία έγκρισης των προϊόντων να την κάνουμε εμείς, ενώ στο μέλλον οι Ηνωμένε Πολιτείε θα κάνουν αυτήν την διαδικασία έγκρισης μέσω τρίτων. Οπότε θα χρειαστεί να διαγράψουμε τις μη ισχύσεις πλέον διατάξεις. Ω συζητητής, χαιρετίζω λοιπόν τις διαπραγματεύσεις και το γεγονός ότι κατέληξαν επιτυχώς ούτως ώστε να έχουμε λοιπόν αυτή τη νέα συμφωνία. Οι τροπολογίες που πρότεινε η Κομισιόν με βρίσκουν σύμφωνο, αλλά μένει ένα ερώτημα ε, ανοιχτό. Διάφοροι κατασκευαστές συμμετέχουν στους δημόσιους διαγωνισμούς μας είπαν ότι συμμετέχουν σε αυτούς τους διαγωνισμούς κυρίως διότι ο εξοπλισμός όπως τον παραγγέλνουν οι αρχές προσαρμόζονται τουλάχιστον ε, στις αρχές και προδιαγραφές του Energy Star. Πιστεύω λοιπόν ότι ο τομέας εφαρμογής ε, του κανονισμού πρέπει να επεκταθεί ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές. Η Κομισιόν δεν ε, ασχολήθηκε με αυτό το θέμα στην πρότασή της, διότι η Κομισιόν πιστεύει ότι οι απαιτήσει για ενεργειακή αποτελεσματικότητα θα προβλέπονται ήδη στην οδηγία για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Όμως, οι διαπραγματεύσεις ε, που γίνονται για αυτήν την οδηγία στο Συμβούλιο νέρωσαν κατά πολύ ε, την ε, ισχύ της οδηγίας αυτής. Πιστεύω λοιπόν ότι θα έπρεπε να προτείνουμε να επεκταθεί το Energy Star ούτω ώστε να μην αφορά μόνο τι κεντρικέ εθνικέ αρχέ, να ισχύει λοιπόν και για τοπικέ και περιφερειακές αρχέ, ούτω ώστε οι παραγωγοί να έχουν περισσότερα κίνδυνα για να συμμετέχουν και σε αυτού του διαγωνισμού. Σα ευχαριστώ πολύ και με χαρά θα ακούσω τώρα την άποψή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον εισηγητή. Δίνουμε το λόγο τώρα στον κύριο Κουκόβιτς που είναι, στην κυρία Κουκόβιτς που είναι Σε Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα σήμερα γιατί πρώτη φορά μας δίνει επεξηγήσεις ο εισηγητής. Στο παρελθόν είχαμε συναντηθεί για να συζητήσουμε αυτό το άκρο σημαντικό θέμα, διότι αφορά τη συμφωνία μεταξύ ΕΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση για ένα συντονισμό των προγραμμάτων επισήμανσης για την ενεργειακή απόδοση. Ως και όδης του ΕΛΚ θα ήθελα να μου γνωμοδοτήσω κι εγώ με τη σειρά μου και να πω ότι είναι η τρίτη παράταση της συμφωνίας μεταξύ ΙΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πρόκειται για αλλαγές ε, τεχνικής υφής, οι οποίες έχουν επέλθει. Δυστυχώς δεν είχαμε πολύ χρόνο να προετοιμαστούμε και να συζητήσουμε το θέμα. Λάβαμε το χρονοδιάγραμμα και προσχέδιο καθώς ε, και τις τροπολογίες δύο εβδομάδες πριν. Εγώ είμαι νέο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ίσως δεν κατανοώ τα πάντα ως προς τα διαδικαστικά ζητήματα, αλλά από τις ε, προηγούμενες από την προηγούμενη μου πείρα ως διαχειρίστρια και πρώην υπουργό, ξέρω ότι το χρονοδιάγραμμα είναι ύψης της σημασίας για να μπορέσουμε να διεκπαιρεώσουμε σημαντικά θέματα. Λάβαμε τροπολογίες από τον εισηγητή και συγκεκριμένα μία και εάν γίνει αποδεκτή τότε οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θα πρέπει να χρησιμοποιούν οπωσδήποτε αυτόν τον κανονισμό, δεσμεύονται δηλαδή. Σε καιρούς κρίσης θεωρούμε ως ΕΛΚ ότι δεν μπορούμε να το προωθήσουμε αυτό. Δεχτήκαμε την οδηγία ενεργειακής αποδοτικότητας πρόσφατα. Προτρέπω όλους να δεχτούν αυτή την οδηγία και να μην ερχόμαστε σε αντίφαση. Στο άρθρο 5 ως προς την οδηγία ενεργειακής απόδοσης, την ε, οδηγία αυτή, αναφέρεται ότι τα κράτη-μέλη θα ενθαρρύνουν τους ε, δημόσιους οργανισμούς σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο να ακολουθήσουν την οδηγία. Νομίζω ότι υπάρχει ασυνέπεια εάν τώρα πούμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους όρους. Εάν λοιπόν η οδηγία ενεργειακής απόδοσης λέει ότι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη, ας αρκεστούμε σε αυτό. Γι' αυτό προτείνω να τροποποιηθεί το κείμενο προτρέποντας τα τοπικά και περιφερειακά ε, όργανα και οργανισμούς καθώς και φορείς να χρησιμοποιήσουν αυτό το πλαίσιο ενεργειακής απόδοσης. Ευχαριστούμε. Η κυρία Χάση έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον εισηγητή μας για την, ε, για την έκθεσή του. Ήμουν ε, η σκιώδη για το προηγούμενο θέμα και συμφωνώ με την βασική προσέγγιση και τις αδερές γραμμές της έκθεσης. Και στην, στον τελευταίο γύρο της συζήτησης είπαμε ότι μόνο ο δημόσιος τομέας θα πρέπει ε, να έχει τέτοιο γραφειακό ε, εξοπλισμό που να ανταποκρίνεται στα κριτήρια του Energy Star. Στο μεταξύ μάθαμε πόσο σημαντική είναι η ενεργειακή απόδοση για όλους ε, τους στόχους μας του συναφείς με την ε, ενέργεια, δηλαδή την πρόσταση του κλίματος, την ενεργειακή ασφάλεια, τη μείωση της εξάρτησής μας από εισαγόμενη ενέργεια. Η ενεργειακή απόδοση λοιπόν είναι κέριο σημείο νευραλγικής σημασίας για την υλοποίηση όλων αυτών των στόχων. Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τις πολιτικές μας, όχι μόνο μέσω της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση, αλλά και με άλλους μηχανισμούς και τρόπους, ώστε οι δημόσιοι διαγωνισμοί και οι δημόσιοι φορείς ε, να εφαρμόσουν και αυτοί με τα προγραμματά τους στους στόχους της ενεργειακής μας πολιτικής. Οι δημόσιοι φορείς ε, είναι κατεξοχήν αγοραστές ε, τέτοιων εξοπλισμών και γι' αυτό μπορεί να αλλάξουν και τους όρους του παιχνιδιού. Άκουσα ε, όταν ξεκίνησε η εφαρμογή του προγράμματος Energy Stars στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θυμάμαι αν ήταν ακριβώς τότε, πάντως άκουσα ότι επί Προεδρίας Κλίντον η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση ε, αποφάσισε ότι από ένα σημείο και μετά θα αγόραζε υπολογιστές ε, μόνο εφόσον πληρούσαν κάποιου στόχου ενεργειακή απόδοση. Και αυτό άλλαξε άρτην ολόκληρο το, το δημόσιο τομέα. Γιατί ακριβώς οι κυβερνητικέ αρχές ήταν ε, κατεξοχήν πελάτης και αγοραστής τέτοιων, τέτοιου εξοπλισμού γραφείου. Οπότε ενισχύουμε την πολιτική μα και αυτή η υποχρέωση ισχύει αυτή τη στιγμή μόνο για τι κυβερνητικέ αρχέ, για τι κεντρικέ κυβερνήσει και μόνο για δημοπρασίε και διαγωνισμού που ξεπερνούν το όριο των 137.000 ευρώ. Οπότε θα πρέπει να λάβουμε κάποια μέτρα για να προωθήσουμε και μια αλλαγή νοοτροπίας σε ό,τι αφορά τις ε, δημόσιες προμήθειες, τις προμήθειες των ε, δημόσιων φορέων, σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο σε κυβερνητικό. Γιατί παραλαμβάνω, οι δημόσιοι φορείς, ο δημόσιος τομέας είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής τέτοιου εξοπλισμού, οπότε η δική του στάση θα έχει μεγάλο αντίκτυπο σε όλο τον κλάδο. Αν λοιπόν εμείς θεσπίσουμε σαφείς κανόνες για την αγορά και τις ε, δημοπρασίες και τους ε, διαγωνισμούς για την αγορά εξοπλισμού γραφείου που θα πληρεί τις προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης, τότε όσοι ασχολούνται με δημόσιες προμήθειες, όχι μόνο σε επίπεδο κυβερνητικών αργών, αλλά και σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ακόμη και σε μικρές ε, πόλεις, σε μικρούς δήμους και κοινότητες, θα αλλάξουν κάπως την οτροπία τους θα αρχίσουν να ευαισθητοποιούνται και να προσέχουν ιδιαίτερα το θέμα της ενεργειακής απόδοσης. Και το τελικό αποτέλεσμα πιστεύω θα είναι επωφελές και για την ε, οικονομία γενικώ. Γι' αυτό και είμαι υπέρ των προτάσεων του εισηγητού για επέκταση αυτής της υποχρέωσης από τις ε, κυβερνητικές αρχές που ισχύει τώρα για όλο το δημόσιο τομέα και για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Επίσης, εγώ θα πρότεινα να καταργηθεί και το όριο αυτό των 137.000 ευρώ. Γιατί συνήθως όταν ο δημόσιος τομέας αγοράζει εκτυπωτές ή υπολογιστές, συνήθως οι αγορές δεν φτάνουν αυτό το όριο, είναι πολύ κάτω από τα 137.000 ευρώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρουμπίκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η συμφωνία μέχρι τώρα ήταν μεγάλη επιτυχία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος είναι λοιπόν να υπάρξουν μέχρι το 2020 εξοικονομήσεις 30%. Η συμφωνία αυτή που εγγράφει το 2000. Αυτό αποδεικνύει ότι η διμερής συνεργασία λειτουργεί σωστά. Η ερώτηση προς την Κομισιόν είναι γιατί μιλάμε μόνο για συνεργασία μεταξύ Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών. Τι προθέσεις έχει η Κομισιόν να συνεργαστεί με την Κίνα, την Ινδία, όπου, όπως ξέρετε, παράγονται, κατασκευάζονται τα περισσότερα ε, τέτοιου τύπου προϊόντα εξοπλισμού Γιατί επίσης να μην λειτουργεί πλέον η, αναγκαία, η αμοιβαία αναγνώριση Υπάρχει καμία δυνατότητα εναρμόνισης. Θα μπορούσαμε να επιδιώξουμε λοιπόν την εναρμόνιση. Δεν θα ήταν ένα θέμα που θα έπρεπε να συζητηθεί σε πολυμερές επίπεδο, ούτω ώστε να έχουμε πλανητικά κριτήρια που να μπορούν και διάφορα Ινστιτούτα για τυποποίηση ή διάφοροι περιφερειακοί οργανισμοί, κοινοβούλια κτλ. να τα εφαρμόζουν. Ευχαριστώ τον κύριο Ρουμπίχ, δεν υπάρχουν άλλοι εγγεγραμμένοι. Γι' αυτό δίνω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Πολ Όντσον. Ευχαριστώ και καλημέρα σας. Συμφωνούμε με τον κύριο Ρουμπίχ και τον εισηγητή ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική συμφωνία έχει επιτελεστεί μεγάλη πρόοδος και έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την ε, ενεργειακή απόδοση διεθνώς. Γι' αυτό συμφωνούμε στην προέκταση της συμφωνίας, στην παράτασή της. Ως προς τη διμερή συνεργασία ΙΠΑ Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είπε και ο κύριος Ρούμπιχ, υπάρχουν πολλά περιθώρια διεθνούς συνεργασίας. Έχουμε ε, συνεργαστεί και με τους Ρώσους, με τους Κίνους, είχαμε συνομιλίες δηλαδή, μέσα στα πλαίσια της διεθνούς ε, δικαιοδοσίας, γιατί θεωρούμε ότι οι ιδέες μας λαμβάνονται υπόψη και από τη Ρωσία και από την Κίνα. Τώρα θα θέλαμε να λάβουμε υπόψη, να ανακτήσουμε δυνάμεις, γιατί έχουμε μείνει αρκετά πίσω μέσα στα πλαίσια του eco-design και ελπίζω να μπορέσουμε να το προωθήσουμε και μέσα στα πλαίσια άλλων δικαιοδοσιών διεθνώς. Δεχόμαστε την προσέγγιση του εισηγητή και αυτό δεν εκπλήσει, γιατί αυτή ήταν και η αρχική μας πρόταση στην Οδηγία Ενεργειακής Απόδοσης. Αυτού λεχθέντος και επειδή βρισκόμαστε στο σημείο έγκρισης της οδηγίας ενεργειακής απόδοσης, βλέπουμε ότι ισχύουν οι ίδιοι όροι μεταξύ κυβερνήσεων και NG Star και θεωρούμε ότι σκοπιμότερο θα ήταν να εφαρμοστεί αυτό το πλαίσιο παρά να παρατείνουμε τις συζητήσεις για το κατά πόσο θα πρέπει να υπάρχει ένα ειδικό και διαφορετικό καθεστώς για τον εξοπλισμό γραφείου από άλλες μονάδες, σε σχέση με άλλες μονάδες παραγωγής και εξοπλισμού. Νομίζω ότι η, ο κύριος Κούκοβιτς, η κυρία Κούκοβιτς είπε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λάβουν υπόψη το επιπρόσθετο κόστος που ενδεχομένως ε, ενέχεται και σε αυτό το στάδιο δεν θεωρούμε ότι θα πρέπει να επεκτείνουμε το πλαίσιο στις τοπικές κυβερνήσεις, διότι θα έχουμε μία αναθεώρηση των δημοσίων συμβάσεων το 2015. Άρα θα επανέλθουμε στο θέμα σύντομα. Ευχαριστούμε την Επίτροπη. Το λόγο έχει ο εισηγητής, ο κύριος Κόβατς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φυσικά και θα λάβουμε υπόψη όλες αυτές τις παρατηρήσεις και θα λάβω υπόψη και τις τροπολογίες όταν τις εξετάσω. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών λοιπόν 16 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας. Περνάμε τώρα στο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης που αφορά την ασφάλεια των δραστηριοτήτων γεώτρησης και παραγωγής φυσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου ανοιχτής θάλασσας. Ο κύριος Ιβο Μπέλετ, ο εισηγητής, έχει το λόγο. Συγγνώμη. Ευχαριστώ για το λόγο. Καλημέρα σας. Αγαπητοί συνάδελφοι, μια και από χθε ξανάρχισε η Νορβηγία της ε, δραστηριότητας γεώτρησης, μπορούμε και εμείς να συνεχίσουμε ε, και τις δικές μας εργασίες για την ασφάλεια σε υπεράκτης πλατφόρμες. Πάνε δύο χρόνια ε, μετά το περιστατικό του Μακάντο στον κόλπο του Μεξικού και την πετρελαιοκυλίδα που ε, ξεκίνησε τη διαδικασία αναθεώρησης της όλης της διαδικασίας που ελπίζουμε ότι θα ολοκληρώσουμε στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας μέχρι το τέλος του έτους αν όλα πάνε καλά. Το σχέδιο εκθεσισμού επί της προτάσεως Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, το έχετε λάβει. Μάλιστα έχει μεταφραστεί και σε όλες τις γλώσσες. Οπότε θα ήθελα επιλεκτικά να αναφερθώ στις αδρές γραμμές της έκθεσης και στις προτινόμενες τροπολογίες. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά τη νομική μορφή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, κατέθεσε πρόταση κανονισμού. Και ο κανονισμός φυσικά έχει το πλεονέκτημα της ε, άμεσης ισχύω και δημιουργεί ένα ομοιόμορφο πεδίο δράσης Προέκυψαν όμως ε, ερωτήματα και προβληματισμό και από τους συναδέλφους και από ενδιαφερόμενου ότι μια τέτοια νομική μορφή του κανονισμού θα δημιουργήσει ένα άλλο επίπεδο ε, νομοθετικό υπεράνω του εθνικού και υπάρχουν φόβοι ότι θα πρέπει να διατυπωθούν οι εθνικές νομοθεσίες οπότε οι ελάχιστοι πόροι ε, από την ε, ασφάλεια θα μετατραπούν σε αυτή την προσπάθεια αναθεώρησης της ε, εθνικής νομοθεσίας, κάτι που θα υποβαθμίσει κάπως τις προσπάθειες για την ασφάλεια. Αυτή ήταν οι φόβοι που διατυπώθηκαν. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο γνωρίζουμε ότι είναι επίμαχο το θέμα. Υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Προτιμούμε όμως αλλαγή της νομικής μορφής και αντί για κανονισμό να έχουμε ένα σαφέ νομικό πλαίσιο, αλλά με τη μορφή οδηγίας. Αυτό προβλέπει η τροπολογία 1. Δεύτερο σημαντικό θέμα και επίσης κέριο αφορά την ανεξαρτησία των αρχών. Ένα από τα βασικά ε, διδάγματα του περιστατικού Μακάντο ήταν ε, η, εξασφάλιση, η σημασία της εξασφάλισης ανεξαρτησίας των ε, αρχών που αφενός αξιολογούν την ασφάλεια και τον, τους περιβαλλοντικούς κινδύνους ε, του εγχειρήματο. Και αυτές οι αρχές θα πρέπει να είναι 100% ανεξάρτητες από τις ε, άλλες αρχές ε, ή τις διοικήσεις που είναι αρμόδιες για την αδειοδότηση των γεωτρήσεων. Φαντάζομαι αυτό το σημείο θα απαιτήσει περαιτέρω διευκρίνηση και εξέταση, γιατί είναι από τα πιο επίμαχα και στο Συμβούλιο. Βέβαια, το Συμβούλιο είναι κάπω πιο προχωρημένο από εμά. Ε, σε εμά θα πρέπει να διευκρινιστούν κάποια ζητήματα αρμοδιότητα. Πάντω και αυτό το θέμα τη ανεξαρτησία των ε, αρχών είναι σημαντικό κεφαλαιόδου σημασία για την περίπτωση αυτή. Τρίτο θέμα, η ανάμεξη του, της ομάδας για την υπεράκτη ασφάλεια. Μια, μια σχετικά νέα ομάδα, αρχές υποπτίας υπεράκτη δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης και τασμάτων πετρελαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια σχετικά νεοπαγής ομάδα. Ε, ξεκίνησε από την έκθεση και το ψήφισμα Ford και με βάση αυτή την έκθεση πέρυσι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο με συντηρητική πλειοψηφία ε, θεσπίσαμε αυτή την αρχή για να αντιμετωπίσουμε τις ε, προκλήσεις από την ασφάλεια σε τέτοιες υπεράκτης πλατφόρμες γεώτρησης και πιστεύω ότι θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος αυτής της ομάδας. Και αυτή ε, η ομάδα αρχών εποπτείας των υπεράκτων δραστηριοτήτων πιστεύω ότι είναι το, ο κατάλληλο μηχανισμός και θα πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως και να διαδραματίσει ρόλος σημαντικός ό,τι αφορά την εφαρμογή του ενωσιακού και των εθνικών πλαισίων. Επίσης λάβαμε υπόψη τη διευρυμένη εντολή του Ευρωπαϊκού, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, του ΕΜΣΑ. Αν ευσταθούν οι πληροφορίες μου, το Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών έχει συμφωνήσει για το νέο πεδίο εφαρμογή του οργανισμού ΕΜΣΑ, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, αλλά έχουμε να ψηφίσουμε και στην Ολομέλεια το θέμα αυτό το Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο. Πάντως είμαι πεπισμένο για την αναγκαιότητα της διευρυμένη εντολή του ΕΜΣΑ, που θα πρέπει να περιληφθεί στα σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και να ξεκινήσουν περιοδικές ασκήσεις για τη δοκιμή των διασυνοριακών μηχανισμών αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Άλλο σημαντικό θέμα είναι η επαλήθευση από τρίτο μέρος. Είναι σημαντικό αυτό το θέμα της επαλήθευσης. Στην, στην έκθεση ε, Ford επισημάναμε την ανάγκη της επαλήθευσης από τρίτο, μέρο. από τρίτο μέρος. Ε, το Συμβούλιο τώρα αφαίρεσε αυτή την έννοια του τρίτου μέρους, γιατί ιδιαίτερα στις μεγάλες εταιρείες έχουμε μια εσωτερική ουσιαστικά επαλήθευση που είναι μια δόκιμη εναλλακτική λύση. Οπότε, στο μέτρο που εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία της, του ελεγκτή, δεν υπάρχει αντίρρηση να γίνεται κατά ανάγκη επαλήθευση από το τρίτο μέρος, αρκεί να είναι ο ελεγκτής ανεξάρτητος το θέμα της ανεξαρτησίας είναι το πλέον σημαντικό εδώ για τη διενέργεια της επαλήθευσης του ελέγχου. Να πω και δύο λόγια για τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις διεθνείς δραστηριότητες, γιατί η οδηγία αυτή φυσικά αφορά το κοινοτικό πλαίσιο, το ενωσιακό πλαίσιο, αλλά υπάρχει μια προφανής προσδοκία και για τους ενδιαφερόμενους, για τις εταιρείε με βάση την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, που ασχολούνται με υπεράκτες δραστηριότητες να ζητηθούν να δραστηριοποιηθούν διεθνώς, σύμφωνα όμως με τα πρότυπα ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε τροποποίησαμε το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να λάβουμε υπόψη αυτή την ανάγκη για τις διεθνείς δραστηριότητες ε, και τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η λογοδοσία, η ευθύνη Προς το παρόν, η, η πρόταση κανονισμού αφορά μόνο την περιβαλλοντική ευθύνη. Υπάρχουν όμως και άλλες μορφές ευθύνης, αστική ευθύνη για παράδειγμα, για ζημίες που εμπίπτουν στο αστικό δίκαιο και μπορούν να απορρέουν από, τέτοιες, τέτοια περιστατικά. Θα πρέπει όλες οι υπεράκτε τέτοιε εταιρείε να καλύπτουν όλο το κόστο των ζημιών από τέτοια ατυχήματα και θα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί χρηματοπιστωτικοί για να καλύπτονται τέτοιου είδου ζημιέ. Αυτέ είναι οι προτάσει μα, δεν είναι καινοφανεί. Υπάρχουν ήδη τέτοια μοντέλα. Προτείνουμε την σύσταση ενό αμοιβαίου σχεδίου αποζημίωση. Νομίζω ότι αυτή ήταν καλή λύση και θα μπορούσε να οργανωθεί σε περιφερειακό επίπεδο. Δεν χρειάζεται ένα πανευρωπαϊκό μοντέλο. Θα μπορούσαμε να έχουμε περιφερειακά μοντέλα ανάλογα με τις περιφερειακές ιδιαιτερότητες. Και φυσικά υπάρχουν και άλλα έκρεμη ζητήματα. Φυσικά δεν είμαστε η μοναδική αρμόδιοι κυρίαρχοι του παιχνιδιού στο θέμα αυτό γιατί και η Νομική Επιτροπή και η Επιτροπή Περιβάλλοντος έχουν κάποιες αρμοδιότητες για το θέμα αυτό. Θα εξετάσουμε φυσικά και τις δικές τους προτάσεις. Ίσως οι δύο επιτροπές ε, έχουν πιο ταχύς ρυθμούς. Εμείς έχουμε αρχές Σεπτεμβρίου την ε, καταληκτική διορία για την υποβολή των τροπολογιών, ενώ οι άλλε δύο τροπολογίε έχουν την επόμενη εβδομάδα ω προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Οπότε έχουν ένα πιο στενόχρονο διάγραμμα από εμά. Αυτή ήταν μια σύντομη επισκόπηση, κυρία Πρόεδρε, των αδρών γραμμών. Επαναλαμβάνω, έκανα μια επιλεκτική παρουσίαση των πιο σημαντικών τροπολογιών και περιμένω τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον εισηγητή. Η κυρία Φόρντ είναι παρούσα. Από ό,τι βλέπω από τους σκιώδεις, και βλέπω άλλους, έχετε το λόγο. Συγχαρητήρια, διότι είναι πολύ αποδοτική εργασία μας. Προτρέχουμε και ε, ζητώ συγγνώμη από τον εισηγητή που προέτρεξε σήμερα το πρωί, να τον συγχαρώ καταρχήν για την εξαιρετική του εργασία και σας ευχαριστώ γιατί λάβατε υπόψη τα σχόλιά μας στην οδηγία ενεργειακής απόδοσης. Θα προβάλλω και άλλες τροπολογίες, αλλά νομίζω ότι οι δραστηριότητες, οι δράσεις της Κομισιόν δεν ήταν επαρκείς. Αν λοιπόν θα έχουμε μία οδηγία, θα ήταν σκόπιμο να ακολουθήσουμε την ίδια γλώσσα, να χρησιμοποιήσουμε την ίδια γλώσσα και στο κείμενο. Εξαιρετική λοιπόν η εργασία σας. Καταστήσατε σαφές ποιος είναι υπεύθυνο, τον κάθε υπεύθυνο για το κάθε θέμα. Μετά από το ατύχημα της πλατφόρμας στον κόλπο του Μεξικού. Ξέρουμε λοιπόν ποιος, που αποδίδονται ευθύνε στις ρυθμιστικές αρχές, στην επιχείρηση, ως προς τον έλεγχο από ένα τρίτο μέρος. Εσείς είπατε ότι αυτό είναι ένα από τα θέματα που μας, που μας απασχολούν. Πολλές φορές λοιπόν χρειάζεται επαλήθευση και από ένα δεύτερο και από ένα τρίτο μέρος, από ένα, από ένα μη εμπλεκόμενο, από ένα μη εμπλεκόμενο φορέα. Δηλαδή δεν μιλάμε για τρίτο μέρος πάντα, αλλά πολλές φορές χρειάζεται. Ως προς την προσέγγιση μίζωνος κινδύνου, θεωρώ ότι αυτό που έχει σημασία είναι να επαληθεύσουμε, να δούμε πού έγκυται το σφάλμα και να αποτιμήσουμε κατά πόσο πρέπει να επέλθουν αλλαγές στις πρακτικές μας. Πρόκειται για μία ζωντανή διαδικασία η οποία ακολουθεί τις εργασίες αυτές σε καθημερινή βάση καθημερινή εξελικτική βάση. Ως προς τα παγκόσμια πρότυπα, δεν μπορούμε να δεσμεύσουμε τους ε, ευρωπαϊκούς φορείς να χρησιμοποιήσουν αυτά τα πρότυπα, δεν είναι δεσμευτικά δηλαδή, αλλά μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτή την οδό. Αυτό είναι ένα θέμα που μας απασχόλησε αρκετά. Και στη δική μου έκθεση δηλαδή ίδιας πρωτοβουλίας ως προς την αστική ευθύνη και ποινική ευθύνη με βάση τα ατυχήματα στον τομέα του περιβάλλοντος ή της υγείας. Εδώ θα πρέπει να επιμείνουμε. Πολλοί λένε ότι καλύπτεται το θέμα από τις άλλες οδηγίες. Εγώ δεν το νομίζω. Νομίζω ότι χρειάζεται μία ειδική ρήτρα θα πρέπει να το καταστήσουμε απόλυτα σαφές. Και ξέρω ότι και άλλες επιτροπές ασχολούνται με το κόστος, με τις δαπάνες καθαρισμού. Νομίζω ότι οι επιχειρηματίες, οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να προβάλλουν μόνο τους χρηματικούς πόρους, αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό. Δηλαδή δεν πρέπει να μιλάμε για αστική ευθύνη ως προς την απόδοση, μάλιστα ένα πρόστιμο, ένα χρηματικό ποσό το οποίο θα πρέπει να αποδοθεί. Θα πρέπει να είναι πολύπτυχη η ευθύνη, θα πρέπει να υπάρχουν φυσικοί πόροι, προσωπικοί πόροι, ανθρώπινο δυναμικό για να καλύψει τις ευθύνες. Αυτό, αυτή τη γλώσσα θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και θα πρέπει να δούμε τι κάνουν και οι άλλες επιτροπές. Σας ευχαριστώ πολύ για την εξαιρετική σας εργασία. Ευχαριστούμε την κυρία Φόρντ. Δεν βλέπω άλλους σκιώδεις, παρόντες, δεν υπάρχουν άλλοι εγγεγραμμένοι. Αν λοιπόν δεν ε, ζητεί κανείς το λόγο, θα τον δώσω στην Επιτροπή για να παρέμβει καταρχήν. Είναι παρόν ο εκπρόσωπος της Επιτροπής έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Και τον εισηγητή και την κυρία Φόρντ για τα σχόλιά της στο κείμενο της πρότασης. Η Επιτροπή καλωσορίζει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον και τον ενεργό ρόλο που παίζει το Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό από την αρχή. Καθώς και την έκθεση ε, ιδίας πρωτοβουλίας που εγκρίνατε πέρυσι. Το κείμενο ε, του εισηγητή είναι μια καλή ανάλυση του προβλήματος. Πιστεύουμε συνολικά ότι ε, βελτιώνει κάποια σημεία του κειμένου. Πολύ καλή βάση εργασίας λοιπόν. Όπως ξέρετε, μέσω της πρότασης αυτής προσπαθούμε να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στους κύριους κινδύνους. Δεν θέλουμε να μπούμε σε δευτερεύοντα θέματα, με επαγγελματικές νόσους ενδεχομένως ή επαγγελματικούς κινδύνους που καλύπτονται από άλλα κείμενα. Ποια είναι τώρα λοιπόν τα θεμελιώδη στοιχεία. Ήδη αναφέρθηκε ο εισηγητής ορισμένα από αυτά. Είναι πρώτα απ' όλα η ανεξαρτησία των ε, αρμοδίων αρχών, ζωτική σημασίας. Συμφωνώ, πρέπει να το δούμε περαιτέρω και το Συμβούλιο θα εξετάσει, θα προσπαθήσει να βελτιώσει τις λεπτομέρειες του κειμένου, αλλά φυσικά πρέπει να αποφύγουμε κάθε σύγκρουση συμφερόντων. Είναι σημείο κλειδί αυτό, πολύ καλό που το αναφέρετε κι εσείς. Σαφέστατα. Έλεγχος από τρίτα μέρη. Και γι' αυτό Αρχικά η Επιτροπή επέμενε να είναι σαφέστατη αυτή η κατεύθυνση, αλλά ακούστηκαν και άλλα επιχειρήματα, εφόσον κάποιες εταιρείες είναι αρκετά ισχυρές για να το κάνουν αυτό, άρα και εδώ μπορούμε ενδεχόμενα να τροποποιήσουμε την άποψή μας, αλλά όχι σε όλες τις περιπτώσεις. Τώρα η νομική μορφή είναι πολύ σημαντικό θέμα. Ξέρω ότι υπάρχουν ε, πολύ έντονες απόψεις γι' αυτό και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Αρχικά προτείναμε κανονισμό. Διότι πρόκειται, διότι θέλαμε να είναι άμεσα εφαρμόσιμη στον κλάδο η απόφασή μας, γιατί ο κλάδος δημιουργεί τους κινδύνους, ο κλάδος θα αποκομίσει και τα ωφέλη. Γι' αυτό επιλέξαμε κανονισμό. Αλλά ακούσαμε ότι υπάρχουν και άλλες απόψεις, ότι μια οδηγία θα ήταν πιο σκόπιμη. Η Κομισιόν θα αντιμετωπίσει με πραγματιστικό τρόπο λοιπόν το θέμα της νομικής μορφής. Θα επιχειρήσουμε να βρούμε την ε, καλύτερη λύση. Τέθηκε και το θέμα υπέτειότητας. Ε, το κείμενο, το κείμενο ασχολείται με την περιβαλλοντική υπετιότητα. Η αστική υπετιότητα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δεν ε, το περιλαμβάνουμε ακόμη στην πρότασή μας. Δεν έχουμε επαρκώς ε, εξετάσει το θέμα για να μπορούμε να προτείνουμε λύσεις. Πρέπει να το δουλέψουμε περαιτέρω. Γι' αυτό ακριβώς είναι υποεκπώνηση δύο μελέτες και μας ενδιαφέρει και η πρόταση του εισηγητή για την αποκοινού εξέταση των κινδύνων. Τι άλλο, τίποτα άλλο. Υπάρχουν και άλλα θέματα, αλλά προς το παρόν αυτά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε την Επιτροπή. Δίνουμε το λόγο στον συνάδελφο Μπέλετ για να συνοψίσει. Ευχαριστώ. Θα είμαι λακωνικότατος. Πολύ επικοδομητικές ε, οι παρεμβάσεις που ακούσαμε. Ευχαριστώ θερμά την κυρία Φόρτ. Νομίζω ότι συμφωνώ και με τις 6-7 προτάσεις και παρατηρήσεις σας. Άρα υπάρχει πλήρης σαφήνεια. Θα πρέπει να προσδιοριστεί σαφώς στο θέμα της ευθύνης, στο θέμα του ελέγχου από τρίτο μέρος, όπως είπε και πρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Φυσικά εξαρτάται από τις, περιστα... από τις περιστάσεις, από τις συνθήκες, από το είδος της εταιρεία. Πάντως υπό ιδιαίτερε περιστάσεις ε, μπορούμε να το επιτρέψουμε, αλλά γενικώ θα πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια το θέμα του ελέγχου από τρίτο μέρος. Επαναλαμβάνω, βρίσκεται σε εξελικτική διαδικασία η έκθεση και το θέμα των, της παρουσίας μας παγκοσμίω και των δραστηριοτήτων διεθνώς είναι πολύ ευαίσθητο θέμα. Θέλουμε να δώσουμε ένα μήνυμα, αλλά από νομική άποψη υπάρχουν δυσκολίες. Ευχαριστώ και τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αστική ευθύνη. Το ανέφερε ο κύριος Έλιο διεξάγονται μελέτες για το θέμα αυτό και νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό το θέμα του επιμερισμού του κινδύνου και της ε, κοινή αντιμετώπισης του κινδύνου. Θα μπορούσαμε να βρούμε μια συμφωνία και να συνεννοηθούμε και με τις επιτροπές ε, περιβάλλοντος και νομικών υποθέσεων για το πολύ σημαντικό αυτό θέμα του risk sharing και risk pooling. Επίσης, αναφέρθηκαν και οι πόροι σε ανθρώπινο δυναμικό γιατί για να διεξαχθούν οι προσπάθειες καθαρισμού δεν χρειάζονται μόνο οικονομικοί πόροι αλλά χρειάζονται και άνθρωποι για να φέρουν σε πέρα τέτοιες διαδικασίες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Φόρτ. Ευχαριστώ τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Έλιο για την πολύ επικοδομητική του στάση. Και χαίρομαι για τη διαβεβαίωση ε, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δείξει ρεαλισμό σε ό,τι αφορά τη νομική μορφή αυτής της πρότασης. Ευχαριστώ πολύ και περιμένω τις επικοδομητικές τροπολογίες των συναδέλφων. Ευχαριστούμε τον εισηγητή, τον ε, κύριο Μπέλετ και τώρα είστε ελεύθεροι μέχρι τις 10.30 διότι εξαντλήσαμε την ημερήσια διάταξη. Στις 10.30 προβλέπεται η επίσκεψη του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων της Κύπρου. Στις 11 θα συναντηθούμε με τον Υπουργό Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού και στις 12 θα συναντηθούμε με τον κύριο Ποτόσνικ θα σας πρότεινα να είστε εδώ στις 10 και 25 έτσι ώστε να αρχίσουμε ακριβώς στις 10 και μισή. Και Η υποβολή τροπολογιών μέχρι στις 4 Σεπτεμβρίου 2012 στις 12 το μεσημέρι. Λοιπόν, μισή ώρα διάλειμμα. Διακόπτουμε τη συνεδρίαση.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 Αναλαμβάνονται οι εργασίες μας. Προβελέπεται λοιπόν η επίσκεψη με η ανταλλαγή απόψεων με τον Υπουργό Ευθύμιο Φλουρέντζο, Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσα στα πλαίσια της Προεδρίας του Συμβουλίου. Ο Υπουργός θα παραμείνει μαζί μας για 45 λεπτά στις 11 και 4 προβλέπεται η λήξη της συζήτησης. Θα δώσουμε το λόγο στον Υπουργό και μπορείτε να εγγραφείτε για να υποβάλλετε ερωτήσεις. Καλώς ορίσατε κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρος, καλή σας μέρα. Θέλω καταρχάς να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τη Δανική Προεδρία για την εξαίρετη δουλειά που έχει επιτελέσει και να ευχαριστήσω και την Επιτροπή σας, κυρία Πρόεδρε, και όλους τους Ευρωβουλευτές της Επιτροπής σας για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μας δίνετε να είμαστε σήμερα εδώ. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, κύριοι Αντιπρόεδροι, έντιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή και ιδιαίτερα, ιδιαίτερη χαρά για μένα που βρίσκομαι σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εδώ που οι θεσμοί και οι αρχές της δημοκρατίας εκφράζονται κατά τρόπο υποδειγματικό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους πυλώνες του οικοδομήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνεται να παρουσιάσω ενώπιον της Επιτροπής σας τις προτεραιότητες και τις στοχεύσεις της Κυπριακής Προεδρίας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, της κοινωνίας της πληροφορίας και της ευρωπαϊκής πολιτικής διαστήματος και παράλληλα να ακούσω τις δικές σας θέσεις και απόψεις. Πιστεύω ακράδαντα πως μόνο μέσα από το γόνιμο διάλογο την αλληλοκατανόηση και τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μπορεί να διαμορφωθούν πολιτικές και νομοθετήματα με γνώμενα πάντα μια καλύτερη Ευρώπη που να ικανοποιεί τις εύλογες προσδοκίες της κοινωνίας των πολιτών. Το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη αποτελεί ένα από τους ακρογωνιαίους λίθους στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Η ανάπτυξη της επόμενης γενιάς ευρυζωνικής υποδομής και η υποστήριξη υποδομών ψηφιακής εξυπηρέτησης αναμφίβολα θα αυξήσουν τις επενδύσεις σε δίχτυα υψηλής ταχύτητας συμβάλλοντας ουσιαστικά στο να ανακτηθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αυξηθεί τόσο η παραγωγικότητα όσο και η καινοτομία. Στο πλαίσιο αυτό, οι διαπραγματεύσεις για την διευκόλυση συνδέοντας την Ευρώπη θα αποτελέσουν προτεραιότητα για την Κυπριακή Προεδρία. Την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο κατά τη Σύνοδο της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού του Ευρωκοινοβουλίου. Οι πρόεδροι του Ευρωκοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Κυπριακής Δημοκρατίας σε κοινή τους δήλωση δεσμεύτηκαν για την όσο το δυνατό στενότερη συνεργασία κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας με κοινό στόχο την υιοθέτηση ενός φιλόδοξου πολιοντούς δημοσιονομικού πλαισίου με επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Η διευκόλυση συνδέοντας την Ευρώπη που αποτελεί σημαντική πτυχή του υποδιαμόρφωση πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου δεν μπορεί να αποτελέσει εξαίρεση. Συνεπώς θα εργαστούμε με το Ευρωκοινοβούλιο κατά τρόπο επικοδομητικό για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για επίτευξη συμφωνίας σε συνάρτηση πάντα με όλες τις άλλες συνιστώσεις του δημοσιονομικού πλαισίου. Επί η Κυπριακή Προεδρία θα επικεντρωθεί στη συνέχιση της εξέτασης μιας σειράς κατευθυντηρίων γραμμών για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Στο πλαίσιο της διευκόλυνσης συνδέοντας την Ευρώπη. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές αναμένεται να στηρίξουν επενδύσεις σε ταχαία και υπερταχαία ευρυζωνικά δίκτυα και πανευρωπαϊκές ψηφιακές υπηρεσίες. Για την Κυπριακή Προεδρία αναμφίβολα αποτελεί προτεραιότητα το εν λόγω θέμα και συνεπώς θα επιδιώξουμε την υιοθέτηση μερικής γενικής προσέγγισης στο Συμβούλιο Δεκεμβρίου. Η ψηφιακή ενιαία αγορά θα τονωθεί με την εφαρμογή της οδηγίας για την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα που θα εξασφαλίζει μια κοινή προσέγγιση σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαμόρφωση του νέου πλαισίου για την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα, η οποία θα έχει σημαντικό θετικό οικονομικό αντίκτυπο, καθώς αναμένεται να δημιουργήσει νέες επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας, θα προωθηθεί σε μεγάλο βαθμό από την Κυπριακή Προεδρία. Εκφράζουμε πλήρη ετοιμότητα να συνεργαστούμε στενά με την Επιτροπή σας για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις επίτευξης συμφωνίας σε πρώτη ανάγνωση. Η Προεδρία δίνει μεγάλη έμφαση στην ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών και θα συνεχίσει με αποφασιστικότητα και επικοδομητική διάθεση τις εργασίες επί του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών ίσα τόσο εντός του Συμβουλίου όσο και σε συνεργασία με την Επιτροπή σας. Επιπρόσθετα, η Προεδρία δηλώνει ετοιμότητα για να ξεκινήσει τις συζητήσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο. Για την προώθηση της ψηφιακής οικονομίας είναι υψής της σημασίας να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών και των επιχειρήσεων στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Ως εκ τούτου η Προεδρία θα εργαστεί επί της πρότασης για ένα πανευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την εμπιστοσύνη στις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά, ηλεκτρονική ταυτοποίηση και υπογραφή με στόχο να επιτευχθεί σημαντική πρόεδρος, πρόοδος επί του λόγω θέματος μέχρι το τέλος της Προεδρίας. Ο ρόλος των νέων και καινοτόμων τεχνολογιών είναι ιδιαίτερα σημαντικός και κατέχει περίοπτη θέση τόσο στη Λευκή Βίβλο για την πολιτική μεταφορών όσο και στο ψηφιακό θεματολόγιο για, τον, για την Ευρώπη η Κυπριακή Προεδρία στα πλαίσια άτυπης συνάντησης Υπουργών Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών που θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Ιουλίου στη Λευκοσία θα επιδιώξει να αναδείξει το ρόλο της ψηφιακής τεχνολογίας στην αηφόρο ανάπτυξη των μεταφορών. Μέσα από την εν λόγω πρωτοβουλία επιδιώκουμε να αναδείξουμε τη σύζευξη, διασύνδεση δύο κεντρικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ψηφιακού θέματολογίου και της πολιτικής μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασική επιδίωξη της συνάντησης μας θα είναι η υποστήριξη των δύο πιο πάνω πολιτικών διαμέσου της προώθησης, ανάπτυξης και βέλτιστης χρήσης των πληροφοριών του δημόσιου τομέα και των ευφυών συστημάτων μεταφορών σε όλα τα μέσα μεταφορών. Η επιτυχής προώθηση των πάνω αναμφίβολα θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της πολυτροπικότητας στις μεταφορές και στη δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου για ηλεκτρονικό σχεδιασμό της μετάβασης των πολιτών από ένα προορισμό σε άλλο κατά τρόπο αποτελεσματικό. Το αποτέλεσμα της συνάντησης ή τα αποτελέσματα της συνάντησης θα παρουσιαστούν στο Παγκόσμιο Συνέδριο για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών ITS World Congress που θα φιλοξενηθεί στην Αυστρία τον προσεχή Οκτώβριο. Στη συνάντηση θα παραστούν οι δύο αντιπροέδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Συν και Νέλη Κρούς, αρμόδιοι επίτροποι για τις μεταφορές και το ψηφιακό θεματολόγιο αντίστοιχα. Έχουν προσκληθεί επίσης και οι προέδροι των δύο κοινοβουλευτικών επιτροπών Ήτρε και Τραν. Ευελπιστούμε να είστε παρούσα στις 16 και 17 του Ιουλίου. Θεωρούμε την παρουσία του Ευρωκοινοβουλίου στην ελόγω συνάντηση επιβεβλημένη και συνεπώς ευελπιστούμε, επαναλαμβάνω και πάλι κυρία Πρόεδρος, να μας τιμήσετε με την παρουσία σας. Η Ευρώπη χρειάζεται μια αποτελεσματική διαστημική πολιτική που θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να καταλάβει ηγετική θέση παγκοσμίω σε επιλεγμένους στρατηγικούς τομείς πολιτικής. Το διάστημα μπορεί να παράσχει τα εργαλεία για την εξέβρεση λύσεων σε πολλές από τις παγκόσμιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία τον 21ο αιώνα και συνεπώς η Ευρώπη οφείλει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στον συγκεκριμένο τομέα. Η Κυπριακή Προεδρία θα επιδιώξει την υιοθέτηση συμπερασμάτων Συμβουλίου σχετικά με τη διαστημική βιομηχανική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπρόσθετα, η Κυπριακή Προεδρία εκφράζει την ετοιμότητά της να εξετάσει στο Συμβούλιο την νομοθετική πρωτοβουλία που αναμένεται να εκδηλωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Γεωεπισκόπησης GMS e με σκοπό την επίτευξη προόδου σε αυτό το σημαντικό τομέα πολιτικής. Η ανάπτυξη του παγκοσμίου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης GNSS, Έκνος και Γαλιλαίο θα συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης. Οι υπηρεσίες του Γαλιλαίου θα αποφέρουν ωφέλη σε όλο το φάσμα των μέσων μεταφοράς θα δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες μέσω της κινητής τηλεφωνίας και θα ενισχύσουν την ασφάλεια των ανθρώπων και των περιουσιών τους. Η Κυπριακή Προεδρία στη βάση της μερικής γενικής προσέγγισης που έχει επιτύχει η Ιδανική Προεδρία στο πρόσφατο Συμβούλιο Υπουργών του Ιουνίου θα προωθήσει τις εργασίες επί της νομοθετικής πρότασης για τη δημιουργία και τη λειτουργία των ευρωπαϊκών συστημάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης η οποία υπόκειται στις διαπραγματεύσεις για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Εκφράζουμε την πλήρη ετοιμότητα μας να εργαστούμε στενά με την Επιτροπή σας για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για επίτευξη συμφωνίας επί του εν λόγω θέματος. Επιπρόσθετα, η Κυπριακή Προεδρία εκφράζει την ετοιμότητά της να εξετάσει στο Συμβούλιο την νομοθετική πρωτοβουλία που αναμένεται να εκδηλωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την οποία θα επιχειρηθεί η τροποποίηση του υφιστάμενου κανονισμού που διέπει τη λειτουργία του οργανισμού GNSS με σκοπό την παρουσίαση έκθεσης προόδου στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου η Κυπριακή Προεδρία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για επιτυχημένη ολοκλήρωση ή επίτευξη προόδου επί των πιο πάνω νομοθετικών προτάσεων. Βασική προϋπόθεση για επίτευξη του πιο πάνω στόχου είναι η αμοιβαία εποφελής συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όλα τα κράτη-μέλη, αλλά κυρίως με το Ευρωκοινοβούλιο κυρία Πρόεδρε, έντιμα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρώτη φορά. Πρόκειται για μια τεράστια πρόκληση. Με πλήρη επίγνωση της ευθύνη και των δυσκολιών αυτού του μεγάλου εγχειρήματο. θα εργαστούμε σκληρά, με σύνεση, με τριοφροσύνη, διαφάνεια και αντικειμενικότητα για να βάλουμε και εμείς το μικρό μας λιθαράκι στην κοινή προσπάθεια για μια καλύτερη Ευρώπη. Προσβλέπω σε μια εξαιρετική συνεργασία κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας και είμαι στη διάθεσή σας για να επιλύσουμε τυχόν προβλήματα και να επιτύχουμε από κοινού τους φιλόδοξους στόχους που έχουμε θέσει για αποτελεσματική προώθηση του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δώσατε να παρουσιάσουμε τις προτεραιότητες και τις στοχεύσεις της Κυπριακής Προεδρίας. Ως καλός ακροατής είμαι έτοιμος να ακούσω τις δικές σας εκτιμήσεις και απόψεις και να απαντήσω στο μέτρο του δυνατού στα ερωτήματά σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Δίνουμε το λόγο στην κυρία Ντελκαστίγιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας ε, καλωσορίζουμε στην Επιτροπή μας που μεταξύ των αρμοδιοτήτων της βρίσκεται και η τεχνολογία επικοινωνίας και πληροφόρησης. Καλωσορίζω λοιπόν την Κυπριακή Προεδρία και θα ήθελα να σας εγγυηθώ ότι και η ομάδα μου και το ΕΛΚ αλλά και όλες οι άλλες ε, ομάδες πάντα θα επιθυμούμε μια στενή συνεργασία και θα είμαστε πάντα διαθέσιμοι για την εκάστοτε Προεδρία. Θα ήθελα να επιμείνω σε ένα από τα θέμα, θέματα που σας απασχόλησαν είναι ένα θέμα που μας απασχολεί ήδη και θα απασχολήσει και την Κυπριακή Προεδρία καθ' όλη τη διάρκεια της, στα πλαίσια της, ε, των τηλεπικοινωνιών. Αφορά το Connecting Europe, το συνδέοντας την Ευρώπη, το οποίο, στο οποίο αναφερθήκατε και εσείς για την ανταλογή δεδομένων. Θα ήθελα να τονίσω τη σημασία αυτού του μέσου. Είτε πρόκειται για δίκτυα μεταφορών, είτε για ενεργειακά δίκτυα, είτε για τηλεπικοινωνιακά. Υπάρχει ένας αλληλοσυσχετισμός, μία αιτιώδης συνάφεια μεταξύ όλων. Στα πλαίσια των τηλεπικοινωνιών Υπάρχει άμεσος συσχετισμός με τα ενεργειακά δίκτυα. Και εδώ μιλάμε και για τα ευφύ δίκτυα που είναι ύψης της σημασίας για να αποκτήσουμε μεγάλη ενεργειακή αποδοτικότητα. Πρόκειται για τρία δίκτυα που είναι ύψης της σημασίας για την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Είτε για την εσωτερική αγορά της ενέργειας, είτε για την ψηφιακή Ευρώπη, είτε για το εμπόριο γενικότερα. Η ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς, όπως τόνισαν και οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, είναι ουσιώδης, έτσι ώστε να προωθήσουμε μια αναπτυξιακή πολιτική μέσω της μεγαλύτερης ανταγωνιστικότητας στις ευρωπαϊκές οικονομίες. Όλη αυτή η επιχειρηματολογία οδηγεί στη ζωτική σημασία της ανάπτυξης των δικτύων και τη συνδεσιμότητα της Ευρώπης μέσω των δικτύων. Θα ήθελα λοιπόν από το δικό σας τομέα να δείτε αυτά τα ζητήματα των δικτύων και της συνδεσιμότητας κατά τους επερχόμενους μήνες. Ελπίζω να έχουμε μία στενή συνεργασία σε αυτό το θέμα και βεβαίως μία διαρκή συνεργασία κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Η κυρία Τόγια έχει το λόγο. Ευχαριστώ και εγώ εξ ονόματος της ε, ομάδας μου θα ήθελα να σας καλωσορίσω κύριε Υπουργέ μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας για την ανάπτυξη και το μέλλον της Ευρώπης. Σας εύχομαι, εύχομαι να έχουμε μια αγαστή συνεργασία και να προωθήσουμε αυτά τα θέματα σε αυτή την κρίσιμη φάση όπου μιλάμε για τον προγραμματισμό των επερχόμενων ετών. Δηλαδή μέσα στα πλαίσια του προσεχούς επταετούς προγραμματισμού. Μιλήσατε για το δημοσιονομικό πλαίσιο και τις ε, δημοσιονομικές προβλέψεις. Αυτά είναι ύψης της σημασίας για την προώθηση των διαπραγματεύσεων ως προς τα δίκτυα μεταφορών, τα ενεργειακά δίκτυα, τα δίκτυα μεταφοράς δεδομένων και το ευρυζωνικό σύστημα. Εάν θέλουμε πραγματικά να εργαστούμε για την ανάπτυξη και εάν επιθυμούμε αυτά τα μεγάλα σχέδια να προωθηθούν, πολλά από αυτά είναι ευρέως γνωστά, θα πρέπει να δούμε πώς θα το επιτύχουμε μέσα στα πλαίσια της διασύνδεσιμότητας, όπως είπε και η κυρία Καρβάλιου, και τα εφή δίκτυα θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα νέα δημοσιονομικά μέσα. Θα ήθελα λοιπόν μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας να συνεργαστούμε έτσι ώστε σε αυτό το εξάμεινο να μπορέσουμε να προωθήσουμε τις διαπραγματεύσεις ως προς τις δημοσιονομικές προοπτικές. Γιατί χωρίς αυτές δεν θα επέλθει καμία πρόοδος στα δίκτυα αυτά και στη γενικότερη ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία θα οδηγήσει και σε θέσεις απασχόλησης και αυτό είναι ο απότερος στόχος. Θα ήθελα λοιπόν να παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγυς αυτές τις διαπραγματεύσεις. Υπάρχει και μία ομάδα επαφής. Δυστυχώς ε, είδαμε ότι δεν μπορέσαμε να προχωρήσουμε υπό τη Δανική Προεδρία, διότι το Συμβούλιο δεν ήταν ιδιαίτερα εύκαμπτο, ευέλικτο ως προς τη διαθεσιμότητα μέσων. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν και τα ομόλογα έργου. Γνωρίζετε ότι αναθεωρήσαμε τον κανονισμό με βάση τις οδηγίες της Κομισιόν. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να τα καταφέρουμε όσο το δυνατόν καλύτερα μέσα στα πλαίσια των μεταφορών και των δημοσίων έργων. Είμαστε, έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην Κυπριακή Προεδρία. Ευχαριστούμε την Πατρίτσια Τόγια. Ο κύριος Κοζανόφσκι έχει το λόγο. se ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω την Κυπριακή Προεδρία και να εκφράσω την ε, χαρά μου για αυτά που είπατε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των δικτύων πληροφορικής. Γιατί εδώ και πολύ καιρό προβληματιζόμαστε με το πώς θα εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη υποστήριξη και καλύτερη συνεργασία για τα διάφορα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης. Γιατί για το μέλλον θα είναι σημαντική η συμβολή τους στην ανάπτυξη και στην εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ μάλιστα είμαι εισηγητής για ένα πρόγραμμα που αναφέρατε και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μία νέα δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για προγράμματα που απορροφούν τεράστιους δημοσιονομικούς πόρους, ε, περίπου στα 20 εκατομμύρια. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη επίβολη πρωτοβουλία. Και επίσης θα πρέπει να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητά μας στον τομέα αυτό, γιατί ε, έχει τεράστιο δυναμικό και οι τεχνολογικές εξελίξεις θα είναι ραγδαίες. Προσβλέπουμε σε πολύ στενή συνεργασία με την Κυπριακή Προεδρία και επίσης θα ήθελα να εκφράσω την ευχή στη διάρκεια της δικής σας Προεδρίας να προωθήσουμε την αντίστοιχη οδηγία που δείχνει σε ποιο βαθμό μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει την ανάπτυξη και τις εξελίξεις στα θέματα αυτά. Γιατί, επαναλαμβάνω, πρόκειται για ένα τομέα με μεγάλο δυναμισμό και τεράστιο δυναμικό για εξέλιξη. Όπως είπε η κυρία Τόκια, είναι πολύ σημαντικό για μας να αναπτυχθούν αυτά τα δίκτυα πληροφορικής. Θα είναι κέρια η συμβολή τους και στην γενικότερη ανάπτυξη. Τα ενεργειακά δίκτυα επίσης ε, είναι ένα άλλο περίπλοκο από τεχνολογικής άποψης ε, θέμα και θα πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας, ε, να συσπυρώσουμε τις δυνάμεις μας για να επιτύχουμε πρόοδο και στο σημείο αυτό. Γιατί θα είναι δύσκολος ο ρόλος της Προεδρίας, γιατί πρόκειται για πολυσύνθετα περίπλοκα ζητήματα. Μπορεί να υπάρχουν κάποια αρνητικά στοιχεία που να επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητά μας, αλλά θα πρέπει να τα περιορίσουμε ώστε να μην δημιουργήσουν προσκόμματα στην ενιαία αγορά. Πάντως μπορείτε να υπολογίζετε στη δική μας υποστήριξη. Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιώδεις και θα συνεργαστούμε επικοδομητικά με την Κυπριακή Προεδρία, ελπίζοντας ότι θα δώσει ιδιαίτερη προτεραιότητα στα θέματα αυτά και φυσικά στις επενδύσεις για τους δορυφόρους. Η κυρία Νίμπλερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, συνάδελφοι, και από πλευρά μου ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας και εύχομαι απόλυτη επιτυχία στην Κυπριακή Προεδρία για τις προσπάθειες που κάνετε για την προώθηση των θεμάτων. Η ψηφιακή εσωτερική αγορά για μένα, για μα. εδώ και πολλά χρόνια μα απασχολεί αυτό που θέλαμε. Για πολλά χρόνια με συνεργασία της ε, Δανικής Προεδρίας αποφασίστηκε ο κανονισμός για το roaming, την περιαγωγή και η οδηγία για τις συχνότητες έχει προωθηθεί πολύ συγκεκριμένη και αναλυτική δουλειά έχει γίνει λοιπόν τους τελευταίους μήνες αλλά όπως είπατε και εσείς κύριε Υπουργέ υπάρχουν και πολλά άλλα που πρέπει να γίνουν συμφωνώ με αυτό που είπε και ο συνάδελφος το Ζενόφσκι για μας βασικό στοιχείο είναι η ευρυζωνική εξάπλωση σε όλη την Ευρώπη η Κομισιόν ε, προσπαθεί, την υποστηρίζουμε όπου μπορούμε. Έχουν ξεκινήσει η συζήτηση και για τα ε, προγράμματα, για τα ομόλογα έργου και στον τομέα των υποδομών και εδώ σας υποστηρίζουμε και ελπίζουμε κατά την Προεδρία σας να προωθηθούν τα θέματα αυτά. Δύο ερωτήσεις, πολύ συγκεκριμένες. Δεν είναι η δική μας αρμόδια επί της ουσίας για το θέμα αυτό, αλλά είναι δική σας αρμοδιότητα, αυτό που θα θίξω, ε, έχουμε νέες προτάσεις για την προστασία των δεδομένων, ο βασικός κανονισμός. Για τη συνεργασία των δημοσίων αρχών. Μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε σε τι βαθμό μεταξύ των κρατών μελών έχει προχωρήσει η συζήτηση και τι στόχους έχετε για το θέμα αυτό κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Θα ήταν δυνατόν δηλαδή να γίνουν κάποιες βασικές κινήσεις για να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου ή αν δεν θα είναι από τα βασικά σημεία της Προεδρίας σας. Και δεύτερη ερώτηση. Συζητάμε για την ε, ε, πληροφορική νεφών. Το θέμα αυτό θα μπορούσατε να το προωθήσετε. Θα, με ενδιαφέρον θα παρακολουθήσω τις απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ο Βιτόριο Πρόντι έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε, σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την παρουσία σας εδώ. Διαπιστώνω με ικανοποίηση ότι δεσμεύεστε για τα δορυφορικά δίκτυα, ως προς τα δορυφορικά δίκτυα, για τη γεωεπισκόπηση και το Γαλιλαίο. Νομίζω ότι θα πρέπει να δράσουμε γιατί πρόκειται για πραγματικά ευρωπαϊκές υποδομές και τεχνολογίες εχμής, καινοτόμες τεχνολογίες που είναι ζωτική σημασίας για να προωθήσουμε τις πολιτικές μας, ιδιαίτερα ως προς το περιβάλλον, τις τηλεπικοινωνίες και την ενέργεια. Γι' αυτό θα πρέπει να προβούμε σε επενδύσεις εν ευθέτω χρόνο, γιατί αντιμετωπίζουμε οικονομικές δυσχέρειες και θα πρέπει να επενδύσουμε άμεσα στις ευρωπαϊκές υποδομές. Αυτό θα ήταν οι ε, ιδεώδες για να βγούμε και από την οικονομική κρίση που διανύουμε. Βασιζόμαστε λοιπόν στη δική σας δέσμευση έτσι ώστε η γεωεπισκόπηση να ληφθεί πλήρως υπόψη μέσα στα πλαίσια των καινοτόμων δημοσιονομικών μέσων του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ρόλος σας είναι πολύ σημαντικός και θα πρέπει να δούμε επίσης και τα ηλεκτρικά δίκτυα τα οποία θα πρέπει να ενημερωθούν με βάση τις νέες τεχνολογίες, έτσι ώστε να περικόψουμε την κατανάλωση κατά εν τρίτων μέσα στα πλαίσια των μεταφορών και να εξορθολογήσουμε τα ηλεκτρικά δίκτυα έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουμε αυτή την σόρευση ενέργειας και ενεργειακής κατανάλωσης. Πρόκειται για ένα θέμα επίγουσας ανάγκης για τους λόγους που σας προείπα. Πιστεύουμε λοιπόν ότι εσείς στο Συμβούλιο θα αφήσετε αυτό το ευρωπαϊκό αποτύπωμα γιατί πρόκειται για υποδομές που έχουν μεγάλη σημασία για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ως Κατά αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να κατανοηθούν. Ευχαριστούμε τον κύριο Πρόντι. Ο κύριος Σοντή έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε θερμά κύριε Υπουργέ για την ευρωπαϊκή δέσμευση και την προσήλωση που δείχνετε στα ευρωπαϊκά θέματα. Επίσης, για τα ευρωπαϊκά δικτύα τηλεπικοινωνιών θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Ε, έχουμε προβλέψει προθεσμία ε, τροπολογιών για τον κανονισμό Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σε ό,τι αφορά τους προσανατολισμούς για τα ευρωπαϊκά δίκτυα τηλεπικοινωνιών. Ε, ευελπιστούμε ότι θα προχωρήσει και θα διεκπαιρεθεί το θέμα επί της Κυπριακής Προεδρίας ό,τι αφορά το ποσοστό κάλυψης για την ευρυζωνικότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει 50% ε, ένα στόχο κάλυψη τη ευρωζωνικότητα. Βέβαια, αυτό δεν πρόκειται να καθησυχάσει του συμπολίτε μα. Ποια είναι η δική σα προσέγγιση, η αντίδραση δεν πιστεύετε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτε θα πρέπει να έχουν ισότιμη πρόσβαση και να εξυπηρετούνται εξίσου όπου και αν βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια, ώστε να δοθεί ε, η πολιτική όθηση και από το Συμβούλιο και από το Κοινοβούλιο για να υπάρχει αυτή η γενική κάλυψη. Δεύτερον, ω προ τη χρηματοδότηση, γιατί αν προβλέψουμε υποχρεώσει κάλυψη θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και τη χρηματοδότησή του. Από αυτή την άποψη δεν δείχνει και ιδιαίτερη φαντασία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον 20ο αιώνα η χώρα μου έχει χρηματοδοτήσει την ηλεκτροδότηση στην Ήπεθρο με μια μικρή υποχρεωτική σφορά στην κατανάλωση και όλοι οι καταναλωτές χρηματοδοτούσαν υποχρεωτικά τα δίκτυα ηλεκτροδότησης και η εξυπηρέτησή τους μέσα στις 15 χρόνια εξασφαλίστηκε σχεδόν παντού. Πώς βλέπετε αυτή την ιδέα μια υποχρεωτική σφορά στην κατανάλωση πανευρωπαϊκής εφαρμογής που θα συγχρηματοδοτούσε ένα επενδυτικό ταμείο ώστε να μπορούμε με ίδιους πόρους να χρηματοδοτήσουμε τις ευρωπαϊκές υποδομές. Για παράδειγμα τα διευρωπαϊκά δικτύα τηλεπικοινωνιών και ταυτόχρονα θα μπορούσε κάτι τέτοιο να ισχύσει όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι για τα ενεργειακά δίκτυα αλλά και άλλα δίκτυα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Οντί. Δεν υπάρχουν άλλοι εγγεγραμμένοι. Επομένως δίνω το λόγο με μεγάλη χαρά στον Υπουργό. Έχετε το λόγο κύριε Υπουργέ. Το μικρόφωνο σας παρακαλώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους όσοι έχετε απευθύνει τον λόγο για την απλότητα με την οποία προσφέρετε την συνεργασία σας προς την Κυπριακή Προεδρία για να μπορέσει να επιτύχει τους στόχους τους οποίους έχει θέσει είτε αυτοί αναφέρονται στις προτεραιότητες τις οποίες έχει καθορίσει είτε αυτοί αναφέρονται στην στα φαγγέλους της σα ατζέντα η οποία θα πρέπει να προωθηθεί από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια της εξάμηνης Προεδρίας. Έχετε θέση κύριε Κασίλο Βέρα διάφορα θέματα. Πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια και την επικοδομητική σας διάθεση για συνεργασία. Οπωσδήποτε η διασύνδεση συνδέοντας την Ευρώπη είναι ένα άκρο σημαντικό θέμα και αποτελεί γι' αυτό προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας. Ασφαλέστατα υπάρχει διασύνδεση στα δίχτυα των τριών τομέων τα δίχτυα αυτά πρέπει να δημιουργούν τις προϋποθέσεις ανάπτυξης σε έργα με πραγματικά προστιθέμενη αξία που να δημιουργούν και τις προϋποθέσεις για επενδύσεις και από πλευράς του ιδιωτικού τομέα. Είναι ίσως και σε αυτή την κατεύθυνση που έχουν υιοθετηθεί το πιλωτικό πρόγραμμα των ομολόγων έργων γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία θα πριμουλκηθεί αν θέλετε και ο ιδιωτικό τομέα να συνεισφέρει ούτω ώστε τα ποσά χρηματοδότηση να αυξηθούν και να μπορέσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να υπάρχουν αυτές οι τεχνολογικές αναπτύξεις. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι είμαστε πλήρως έτοιμοι για συνεργασία με το Ευρωκοινοβούλιο σε αυτόν τον τομέα. Νομίζω ότι και με την κυρία Τόλα θα συμφωνήσουμε για τη σημαντικότητα των δικτύων μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και ενεργειακής πολιτικής. Θα εργαστούμε όσο το δυνατό καλύτερα και σκληρότερα αν θέλετε, ούτω ώστε αυτοί οι τομεί να έχουν τη σημασία την οποία θα πρέπει να έχουν γιατί αντιλαμβανόμαστε και την σημαντικότητά τους στην ανάπτυξη αλλά και στην κίνηση παραπέρα της τεχνολογικής αναβάθμισης που θα δημιουργήσει συνθήκες ανταγωνιστικότητας στην ευρωπαϊκή οικονομία. Από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεστε ότι και το ΣΕΦ συζητείται μέσα στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου η οποιαδήποτε απόφαση θα ληφθεί θα είναι μετά από τις συζητήσεις οι οποίες θα γίνουν μέσα στο Συμβούλιο θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε όσο το δυνατό καλύτερη πρόοδο και σίγουρα ο στόχος της Κυπριακής Προεδρίας είναι η επίτευξη συμφωνίας σε συνάρτηση πάντα με όλες τις άλλες συνιστώσεις. Όσον αφορά την ερώτηση την οποία, η τοποθέτηση την οποία έχει θέσει ο κύριος Σοζανόσκι για τα δορυφορικά συστήματα είναι χωρίς αφιβολία ένα σημαντικός τομέας που δημιουργεί σημαντικά άμεσα και έμμεσα ωφέλη στην οικονομία της Ευρώπης, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα εργαστούμε για αυτό το θέμα με επίγνωση της σοβαρότητας για να διασφαλίσουμε από κοινού την έγκαιρη εγκατάσταση της εφαρμογής τους. Αντιλαμβανόμαστε πλήρω το πόσο σημαντικά προγράμματα είναι ότι θα πρέπει να εγκατασταθούν το συντομότερο δυνατό για να βάλουν την Ευρώπη σε ανταγωνιστική τροχιά αυτό το οποίο μπορούμε να υποσχεθούμε είναι ότι θα πράξουμε ότι είναι δυνατό από δικής μας πλευράς να κατανοήσουν οι άλλοι φορείς της απόφασης την αναγκαιότητα και το επίγον της λειτουργίας αυτών των προγραμμάτων. όσον αφορά τα ερωτήματα τα οποία έχετε θέσει η κυρία Νίπλερ για την χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα σίγουρα έχει επιτευχθεί μεγάλη πρόοδος στο Συμβούλιο επί της Δανικής Προεδρίας νομίζω ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις μέσα από το διάλογο μαζί σας να έχουμε συμφωνία. Θα όσον αφορά τα θέματα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ασφάλεια του διαδικτύου. Δεν έχει ακόμα εκδοθεί ανακοίνωση, αναμένεται να εκδοθεί τον ε, Σεπτέμβριο. Στόχος μας είναι να υπάρξει ανταλλαγή απόψε στο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών του Δευτέρου, του, του Δεκεμβρίου. Και αυτό έχει να κάνει με την ασφάλεια φυσικά του διαδικτύου, το κύβερνο έγκλημα και την εξωτερική διάσταση των πληροφοριών. Όσον αφορά το cloud computing, ε, είναι σημαντική πρωτοβουλία. Εκφράζουμε την ετοιμότητα να εξετάσουμε την όποια πρόταση θα κατατεθεί από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. έχετε θέσει ή κάνει κύριε πρώτη κάποιες επισημάνσεις για τις οποίες έχετε απόλυτο δίκιο. Πρέπει να κινηθούμε έγκαιρα για να διασφαλίσουμε τις απαραίτητες πιστώσεις όπως έχω πει και προηγουμένως και έχω δώσει την υπόσχεση για να προχωρήσουν τα προγράμματα τα οποία είναι άκρο σημαντικά όπως είναι το GMS. E Βρισκόμαστε εν αναμονή των συζητήσεων για τον προϋπολογισμό και θα κινηθούμε άμεσα να εξετάσουμε την όποια νομοθετική πρωτοβουλία κατατεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. κύριος Όντι θα πρέπει να πω ότι είμαστε έτοιμοι για μερική γενική προσέγγιση στα θέματα των διευρωπαϊκών δικτύων για το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Αντιλαμβανόμαστε και εδώ την σημαντικότητα και θα εργαστούμε σκληρά ούτω ώστε τουλάχιστον να έχουμε αυτή την προσέγγιση τη μερική κατά το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. συμφωνούμε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες όπου και να βρίσκονται. Πρέπει να προωθήσουμε έργα και προτάσεις που θα δημιουργούν αυτές τις προϋποθέσεις και φυσικά όπως έχουμε μπει και προηγουμένως μέσα από τις επενδύσεις και του ιδιωτικού τομέα. Πρέπει μέσα από αυτό το φάσμα της πολιτικής σε όλους τους τομείς. Είτε πρόκειται για τα διευρωπαϊκά δίχτυα τηλεπικοινωνιών, είτε πρόκειται για τα διευρωπαϊκά δίχτυα μεταφορών, είτε πρόκειται για τα άλλα προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης και επισκόπησης της ε, γης, πρέπει να επιτύχουμε την οικονομική, εδαφική και κοινωνική συνοχή της Ευρώπης. Νομίζω ότι θα πρέπει κάθε προεδρία να βάζει το δικό της λιθαράκι προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ για την παρουσία σας και για την διαθεσιμότητά σας. Απαντήσατε σε όλες μας τις ερωτήσεις, δεσμευθήκατε και όπως γνωρίζετε, στην Κύπρο προβλέπεται μία συνάντηση για την ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών. Θα δούμε κατά πόσο μπορεί να μεταβεί κάποιο μέλος της ε, δικής μας Επιτροπής. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ και σας ε, ευχόμαστε καλή επιτυχία. Γεια σας. Παραμένουμε στην αίθουσα γιατί έχει φτάσει ο επόμενος Υπουργός.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 Συνεχίζουμε με την ε, δεύτερη φάση της συνάντησης των συναντήσεών μας. ορίζω τον Υπουργό Νεοκλή Σιλικιώτη, Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσα στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας. Καλώς ορίσατε, κύριε Υπουργέ. Περιμένουμε να ακούσουμε την εισήγησή σας. Έχετε το λόγο. Ε, <clears throat> κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Αντιπρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτές, μέλη της και μέλη της ε, Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ίντρε, κυρίες και κύριοι, η σημερινή παρουσία μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συγκεκριμένα ενώπιον της Επιτροπής Ίντρε δίνει τη συνέχεια στην καθημερινή πρακτική να ενημερώνεστε από την Προεδρία του Συμβουλίου για τι προτεραιότητες και δράσει που αναλαμβάνει να προωθήσει κατά διάρκεια τη εξάμεινη ιδείας στα θέματα βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ενέργεια. Όμω πολύ πέραν τη ανταπόκριση μου σε καθιερωμένες πρακτικέ, η εδώ παρουσία μου είναι δηλωτική πράξη του σεβασμού μου απέναντι στο θεσμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κρίσιμου ρόλου που διαδραματίζει για να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση δημοκρατικότερη, για να πλησιάσει περισσότερο και να φουγκράζεται καλύτερα του πολίτε τη. Άλλωστε, το κεντρικό μήνυμα και βασική προσπάθεια της Κυπριακής Προεδρίας είναι για μια καλύτερη Ευρώπη, πρώτα και κύρια για τους πολίτες της. Από την έναρξη ισχύω τη συνθήκη τη Λισαβόνα έχουν διευρυθεί οι αρμοδίδε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ω συνομοθέτη με το Συμβούλιο. Ω η Προεδρία του Συμβουλίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνουμε την ετοιμότητά μα να συνεργαστούμε στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έτσι ώστε να προωθήσουμε με επιτυχία του φακέλου που θα διαχειριστούμε το δεύτερο εξάμεινο του 2012 στους τομείς της αρμοδιότητάς μας σχετικά με τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και την ενέργεια. Στην αρχική μου αυτή παρέμβαση συνοπτικά θα σας παρουσιάσω τις βασικές μας πολιτικές και τα επιμερούς θέματα που θα διαχειριστούμε κατά τους επόμενους έξι μήνες όπως συμφωνήθηκα στο πλαίσιο του τρίου της Προεδρίας. Με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο την Πολωνική όσο και τη Δανική Προεδρία για τη συνεργασία που αναπτύξαμε όλη αυτή την περίοδο αλλά και να του συγχαρώ για την επιτυχή διαχείριση σημαντικών φαγγέλων που Σε ό,τι αφορά την επιχειρηματικότητα και τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Είναι σημαντικό που η Ευρώπη φαίνεται να πήρε την απόφαση να επιστρέψει και πάλι στην ανάπτυξη. Και ανάπτυξη σημαίνει, μεταξύ άλλων, προώθηση πολιτικών που ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και ειδικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το θέμα αυτό θα αποτελέσει την ναυαρχίδα της Προεδρίας μας στον τομέα της ανταγωνιστικότητας. Η τρέχουσα οικονομική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνο με μέτρα αυστηρής λιτότητας. Απαιτούνται ταυτόχρονα μέτρα ανάπτυξης και στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ως γνωστόν αποτελούν το βασικό κορμό της οικονομίας της Ευρώπης. Εθαρρύνουν την κοινοτομία και δημιουργούν συνθήκε απασχόληση, συμβάλλοντα έτσι στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Στο πλαίσιο αυτό, η Κυπριακή Προεδρία και σε συνέχεια της συμφωνίας που επιτεύχθη κατά το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας στις 30 Μαΐου του 2012 θα προωθήσει την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το πρόγραμμα COSME 2014-2020 και θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για τη σύγκληση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό που προέχει κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο είναι να σταλεί από όλα τα αρμόδια θεσμικά όργανα της Ευρώπης ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα για την ανάγκη ουσιαστικής και άμεσης στήριξης της επιχειρηματικότητας και ειδικότερα και ειδικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αναφυσβήτητα πλήττονται και περισσότερο από την οικονομική κρίση. Προς την κατεύθυνση αυτή θα επικεντρωθούμε παράλληλα στην ανάδειξη τη σημασία τη επιχειρηματικότητα για του νέου ανθρώπου, στην καλλιέργεια επιχειρηματική κουλτούρα από τι νεαρέ ηλικίε, στην ενίσχυση τη επιχειρηματικότητα μεταξύ ειδικών πληθυσμιακών ομάδων, καθώ και στην παροχή δεύτερη ευκαιρία σε έντιμου επιχειρηματίε, <clears throat> οι οποίοι όμω είχαν την ατυχία να βιώσουν μια χρεοκοπία. Υπό τι παρούσε οικονομικέ συνθήκε, η Ευρώπη χρειάζεται μια νέα γενιά επιχειρηματιών οι οποίοι με την κατάλληλη υποστήριξη θα μπορούν να αναπτύσσουν και να μετρησιώνουν τις ιδέες τους σε νέα προϊόντα και υπηρεσίε. Το θέμα της επιχειρηματικότητας θα συζητηθεί διεξοδικά στο άτυπο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας που θα πραγματοποιηθεί στη Λευκοσία στις 18 και 19 Ιουλίου. Παράλληλα με τις ανωτέρω πρωτοβουλίες, έφαση θα δοθεί και στην παρακολουθήση της πορείας εφαρμογής τόσο από τα κράτη-μέλη όσο και από την Επιτροπή της ολοκληρωμένης πράξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τη Small Business Act, μέσω της σχετικής έκθεσης που θα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Κυπριακή Προεδρία θεωρεί πως είναι ιδιαίτερα σημαντικό ακριβώς τέσσερα χρόνια μετά την υιοθέτηση της πρωτοβουλίας Small Business Act για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εξεταστεί η πρόοδος που έχει συντελεστεί και να εντοπιστούν οι δράσεις και οι πολιτικές εκείνες που πρέπει να δυναμωθούν περαιτέρω. Λαμβάνοντα υπόψη όλα τα παραπάνω, στόχο τη Προεδρία τη Κύπρου είναι η υιοθέτηση πολιτικών συμπερασμάτων για την επιχειρηματικότητα από το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητα που θα πραγματοποιηθεί στι 10 Δεκεμβρίου του 2012. Σε ό,τι αφορά τώρα στον τομέα τη ε, βιομηχανική πολιτική. Για τον τομέα τη βιομηχανία, η Κυπριακή Προεδρία θεωρεί ότι είναι επίση κεφαλαίου σημασία για την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία στην Ευρώπη. Η βελτίωση τη ανταγωνιστικότητα τη ευρωπαϊκή βιομηχανία μπορεί να μειώσει το κόστο και τι τιμέ των προϊόντων, να βελτιώσει την ποιότητα και να προωθήσει την καινοτομία, συμβάλλοντα κατά αυτόν τον τρόπο στη δημιουργία νέων θέσεων εργασία και στην αύξηση τη παραγωγικότητα στο σύνολο τη οικονομία. Η μεταπικητική βιομηχανία και οι συναφεί με αυτήν οι υπηρεσίες αντιπροσφεύγουν περισσότερο από το 50% τη απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα, το 75% των εξαγωγών και το 80% των ιδιωτικών επενδύσεων έρευνα και ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην κατεύθυνση αυτή υποστηρίζουμε τη νέα βιομηχανική πολιτική η οποία, η οποία αποτελεί μια από τι 7 εμβληματικέ πρωτοβουλίε τη στρατηγική Ευρώπη 2020 και κατά τη διάρκεια τη Προεδρία μα σκοπεύουμε να εξετάσουμε την επικείμενη ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την επισκόπηση τη πορεία εφαρμογή τη. Η Κυπριακή Προεδρία θεωρεί πω υπό το πρίσμα τη παρούσα οικονομική κατάσταση είναι σημαντικό να εντοπιστούν οι επιμέρου προτεραιότητε τη βιομηχανική πολιτική που πρέπει να ενισχυθούν προτείνοντα κατάλληλε τροποποιήσει ή και βελτιώσει. Επίση, σε τομεακό επίπεδο θα εξεταστεί η πρωτοβουλία για τι πρώτε ύλε, ο τομέα τη αυτοκινητοβιομηχανία, οι βασικέ τεχνολογίε γενική εφαρμογή καθώ και η ναυπηγική βιομηχανία. Σε ό,τι αφορά τον τομέα τη ενέργεια, έχοντα αναφερθεί στι προτεραιότητες μα όσον αφορά τον τομέα τη βιομηχανική πολιτική, να μου επιτρέψετε τώρα να αναφερθώ στι προτεραιότητες μα όσον αφορά στον τομέα τη ενέργεια. Η ασφαλής αηφόρος και οικονομικά ενέργεια, η οποία θα συμβάλλει στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και στην ευφύ βιώσιμη και χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς ανάπτυξη αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρώπη. Η δράση σε ενωσιακό επίπεδο μπορεί να και πρέπει να προσδώσει προστιθέμενη αξία στο στόχο αυτό και η Κυπριακή Προεδρία θα αφοσιωθεί στη συνέχιση του σημαντικού έργου που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα ο εξυγχρονισμός και η ανάπτυξη των ευρωπαϊκών ενεργειακών υποδομών και η διασυνοριακή διασύνδεση των δικτύων είναι ιδιαίτερη σημασία προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και η εκδήλωση αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, η ασφάλεια εφοδιασμού της Ένωσης, καθώς και η πρόθεση της ενεργειακής αποδοτικότητας και της ανάπτυξης νέων και ανανεώσιμων μορφών ενέργεια. Η πρόταση κανονισμού σχετικά με τις κατευθυντήρες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας. Με δεδομένη την ανάγκη για ταχύ ανέναξη συγκεκριμένων έργων, θα συμφωνούσαμε στο στόχο για συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση πριν το τέλος του χρόνου. Κάτι τέτοιο βέβαια θα ήταν εφικτό αν τηρηθούν κάποια σφιχτά χρονοδιαγράμματα Προ αυτήν την κατεύθυνση θα βοηθούσε αν η Ήτρε καταλήξει τι συστολικέ τροπολογίε το συντομότερο δυνατό, τι προτινόμενε τροποποιήσει έτσι που το Συμβούλιο να μπορεί να αρχίσει να τι εξετάσει. Σημαντικό είναι επίση για να προλάβουμε τα χρονοδιαγράμματα είναι να μην υπάρξουν καθυστερήσει που θα οφείλονται στι παράλληλε συζητήσει επί του νέου πολιετέ δημοσιονομικού πλαισίου και τη διευκόλυνση συνδέοντα την Ευρώπη. Ευθύνη όλων μα είναι να παραδώσουμε έγκαιρα τους κανόνες και το ρυθμιστικό πλαίσιο που θα διέπει την ανάπτυξη των ενεργειακών υποδομών ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και να διασφαλίσουμε την επίτευξη των στόχων που από κοινού έχουμε θέσει για 20% μείωση των εκπομπών αερίου θερμοκηπίου, 20% αύξηση του μεριδίου των ανάσιμων πηγών ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας και αύξηση του ε, ποσοστού ενεργειακής απόδοση σε 20%. Η Ένωση έχει συμφέρον να διατηρήσει την εχώρια παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου για λόγου ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, καθώ και για τη διατήρηση των θέσεων εργασία και των επιχειρηματικών ευκαιριών τη ευρωπαϊκή οικονομία. Παρά το γεγονό ότι δεν είναι δυνατή η πλήρη εξάλληψη των κινδύνων από τι περισσότερε ανθρώπινε δραστηριότητε, συμπεριλαμβανομένου και του κλάδου των υπεράχτιων δραστηριοτήτων υδρογοναθράκων, θα πρέπει να κατοχυρώνεται η ασφάλεια και η ακυρότητα των εργασιών και η μέγιστη προστασία των Ευρωπαίων πολιτών και του περιβάλλοντος. Η Κυπριακή Προεδρία έχει θέσει τον προτινόμενο κανονισμό για την ασφάλεια των υπεράκτιων δραστηριοτήτων αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου στις προτεραιότητες της. Θα επιδιώξουμε πρόοδο στις ειδήσεις εντός του Συμβουλίου καθώς και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπου η έναρξη των διαπραγματεύσεων διαφαίνεται εφικτή. Ενημερωτικά να προσθέσω πως το θέμα αυτό όπως και η ασφάλεια της ενεργειακής τροφοδοσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης υπουργικής διάσκεψης που διοργανώνουμε στην Κύπρο στις 9 Νοεμβρίου σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη συμμετοχή των κρατών μελών και των χωρών της Νοτανοητική Μεσογείου. Η Μεσόγειος, όπως γνωρίζουμε, είναι μια κλειστή θάλασσα. Συνεπώς, για να την προστατεύσουμε δεν αρκεί τα μέτρα που θα λάβουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται να υπάρξουν σύμφωνα συνεργασίας με τους γείτονές μας και στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου βρίσκεται σε εξέλιξη ερευνητικέ, ερευνητικές αλλά και άλλες γεωτρήσεις και χρειάζεται ακριβώς να καταλήξουμε σε συμφωνία με τους γείτονές μας. Θα πρέπει σε αυτή την προσπάθεια να εμπλέξουμε και, του, ε, και τους γείτονές μας. Είναι με αυτό το σκεφτικό που θέλουμε μέσα από αυτή τη ε, διάσκεψη να καταλήξουμε σε μία κοινή διακήρυξη που θα πρέπει να εφαρμόζουν όλες οι χώρες για τον περιορισμό των κινδύνων και των ατυχημάτων, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντο όταν επιχειρούνται υπεράχτιε δραστηριότητε αναζήτηση ή εκμετάλλευση υδροναθράκων. Περνώντα σε ένα άλλο θέμα, σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η Κυπριακή Προεδρία έχει ως στόχο την υιοθέτηση συμπερασμάτων του Συμβουλίου τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Πιστεύουμε ότι η περαιτέρω αύξηση της συνεισφοράς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απαιτεί παράλληλες πολιτικές όπως την πρόθεση των κατάλληλων υποδομών και διασυνδέσεων και την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, στόχο μα είναι να λάβουμε επίση υπόψη τι κατευθύνσει που έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω τη ανακοίνωσή τη για τον ενεργειακό χάρτη πορεία 2050. Για τον χρονικό ορίζοντα πέραν του 2020, η ανακοίνωση αναγνωρίζει ότι χωρί κατάλληλο πλαίσιο η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια θα επιβραβευθεί. Κάτι το οποίο συμμεριζόμαστε κι εμεί. Ω εκ τούτου, προτείνουμε να ξεκινήσει η διαδικασία για την προετοιμασία μελλοντικών επιλογών πολιτικής και οροσίμων για το 2030. Λόγω της σημασίας του θέματος, όχι μόνο για το Συμβούλιο αλλά και για το Κοινοβούλιο, έχουμε αποστείλει προσκλήσεις για συμμετοχή και ως συζητητών Ευρωβουλευτών στην άτυπη συνάντηση Υπουργών που θα έχουμε στις 17 Σεπτεμβρίου στην Κύπρο, που κύριο θέμα στην ατζέντα θα είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επίσης, κατά τη διάρκεια της εξάμηνης μας Προεδρίας, προσδοκούμε στην επίτευξη συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί της πρότασης κανονισμού για το πρόγραμμα επισήμασης της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου, την Energy Star. Πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα Energy Star, το οποίο ακολουθεί μια συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου 20% εξοικονόμησης ενέργειας μέχρι το 2020. Παράλληλα, βέβαια, μια σύντομη κατάληξη επί αυτού του θέματο θα έκλεινε το νομικό κενό που παρατηρείται δεδομένου ότι η τρέχουσα συμφωνία έχει λήξει. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ. Έχω δέκα εγγεγραμμένους. Γι' αυτό θα ήθελα να περιοριστείτε κάπως για να μπορέσει να μας απαντήσει ο Υπουργός. Ο κύριος Καντσάν. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, για την παρουσία σας και για την εισήγησή σας. Νομίζω ότι τα δύο μεγάλα θέματα που αφορούν ε, την ενέργεια και τη βιομηχανία ενστερνίζονται την έννοια της ανταγωνιστικότητας. Αυτό είναι το θεμελιώδες στοιχείο το οποίο δεν θα πρέπει να παραλείψουμε. Γιατί σήμερα ζούμε σε μια Ευρώπη η οποία δεν είναι ανταγωνιστική. Άρα δεν είμαστε σε θέση να προωθήσουμε μια σωστή δράση ενδοκινοτικά και εξοκινοτικά. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να τονίσουμε την τεχνογνωσία και την καινοτομία. Γιατί όταν μιλάμε για ΜΜΕ γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να διαθέτουν την τεχνογνωσία και να μπορούν να δρουν συλλογικά. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να σταθούμε σε αυτό το στοιχείο. Ως προς τον τομέα της ενέργειας, δεν άκουσα να μας πείτε κάτι για την πυρηνική ενέργεια. Δεν ξέρω κατά πόσο θεωρείτε ότι πρόκειται για μια επικίνδυνη μορφή ενέργειας ή όχι. Πώς τη βλέπετε στο πρόγραμμά σας. Ως προς τον ενεργειακό τομέα γενικότερα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι συσχετίζεται με την απασχόληση και με την κοινωνική συνοχή. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ανταγωνιστικότητα και επικαιροποίηση των δεδομένων. Επίσης, δεν αναφερθήκαμε σε θέματα χρονισμού και πόρων. Δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το πρόγραμμα συνδέοντας την Ευρώπη ή κατά πόσο θα πρέπει να εξεύρουμε άλλες αγορές κεφαλαίων. Κύριε Υπουργέ, ο προγραμματισμός 14-20 30-50 καλώς βαίνει, αλλά θα πρέπει να προβάλλουμε άμεσες πρωτοβουλίες που να δώσουν αμεσότερα καρπούς. Θα πρέπει λοιπόν να επινοήσουμε μία βραχυχρόνια πολιτική για να αντιμετωπίσουμε και αυτό το μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα που υφίσταται στην Ευρώπη. Van Brent. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Είχαμε ήδη την ευκαιρία να σας συναντήσουμε στην πανέμορφη, ηλιόλουστη και ζεστή σας πατρίδα. Δεν θα επαναλάβω τα συμπεράσματα των συναδέλφων, αλλά διαπιστώσαμε ότι η Κυπριακή Προεδρία έχει όλα τα ατού στα χέρια της για να γίνει μια εξαιρετική Προεδρία. Εγώ είμαι Βελγίδα, κατάγομαι και εγώ από μικρή χώρα και διαπιστώνουμε ότι στις μικρές χώρες, επειδή ακριβώς τα εθνικά συμφέροντα είναι πιο μικρά, οι μικρές χώρες είναι πιο διαλλακτικές και πιο διατεθειμένες για την ανέβρεση συμβιβαστικών λύσεων. Μας ε, εκθέσατε τα πιο κατεπήγοντα οριζόντια θέματα που θα σας απασχολήσουν, τα ζητήματα της ενέργειας, της μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τη επιχειρηματικότητα. Μιλήσατε όμως και για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Γνωρίζω ότι η φιλοδοξία σας είναι να καταλήξετε σε συμφωνία στο Συμβούλιο για το θέμα αυτό και σας εύχομαι ολόψυχα καλή τύχη. Πάντως, συμφωνούμε προς ένα σημείο. Χρειαζόμαστε ένα φιλόδοξο ε, χρηματοδοτικό πλαίσιο ε, και επενδύσεις φυσικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μην μιλάμε μόνο για οικονομίες, για εξοικονόμηση, αλλά και για επενδύσεις. Θα ήθελα να σας θέσω μία ερώτηση. Ο χάρτης πορείας, ο δικός χάρτης ε, για το 2050 και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εμείς ε, στην ομάδα μου, δεν είμαστε οι μόνοι άλλωστε, θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να καταλήξουμε σε συμφωνία και να αναζητήσουμε μια συμβαστική λύση για να υπάρξουν δεσμευτικοί ε, στόχοι σε ό,τι αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση και τη μείωση των καυσαερίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το περίφημο τριπλό 20 γιατί να μην είμαστε πιο φιλόδοξοι, να το κάνουμε 30, 40, 50. Είναι πιο φιλόδοξο, αλλά αν θέλουμε στόχους για το 2050, νομίζω ότι οι στόχοι 30, 40, 50 είναι πιο δόκιμοι. Δεν ήθελα να αναφερθώ στην πυρηνική ενέργεια, αλλά μια και το έθιξε ο κύριος Καντσιάν, δεν μπορώ να σιωπήσω. Το συζητήσαμε ε, στην Κύπρο με κάποιους ευρωβουλευτές. Πολλοί ε, ε, αντέδρασαν στην Κύπρο για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν διαμαρτυρήθηκε και δεν αντέδρασε σε ό,τι αφορά το σχέδιο κατασκευής πυρηνικού σταθμού στην Τουρκία. Όπως ξέρετε, η πυρηνική ενέργεια θεωρείται τόσο ασφαλές μέσω ενέργειας που πολύ συχνά κατασκευάζονται πυρηνικοί αντιδραστήρες κοντά στα σύνορα με άλλες χώρες, κάτι που de facto δημιουργεί απειλή για τις γειτονικέ χώρες. Εσείς τι περιμένετε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προσδοκάτε μια σχετική πρωτοβουλία. Ευχαριστώ και παραλαμβάνω καλή τύχη στην Κυπριακή Προεδρία. Grazie, il collega Ευχαριστώ πολύ. Ρόδε, please. Ρόντε. Ο κύριος Ρόντε έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Και σας ευχαριστώ για την πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία και τους στόχους που μας παρουσιάσατε. Χαιρόμαστε ιδιαίτερος και νομίζω ότι είναι ευάρεστο που εστερνιζόμαστε πολλούς στόχους τα τρία θεσμικά όργανα. Αυτό που λείπει από αυτά που ακούσαμε είναι κάτι που συχνά επισημαίνω στις διαδοχικές προεδρίες. Αυτό που λείπει λοιπόν είναι η απάντηση ε, στην ερώτηση πώς θα τα καταφέρουμε όλα αυτά. Γιατί ωραία είναι τα συνθήματα, πολύ δημοφιλή, ανάπτυξη κτλ. Το θέμα είναι πώς θα τα υλοποιήσουμε, πώς θα καταλήξουμε σε αυτά αποτελέσματα για αυτές τις ε, θεάρεστες δηλώσεις που κάνουμε. Για να σας βοηθήσω λοιπόν θα υποβάλω μια πλούστατη πρόταση για να εξασφαλίσουμε την πραγμάτωση αυτών των ε, πολύ ωραίων προθέσεων και στόχων για να αποφύγουμε τα σφάλματα των προηγούμενων προ... προεδριών, δηλαδή να δημιουργήσουμε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο με πολλές αγαθές προθέσεις αλλά ελάχιστα έργα, είναι να δώσουμε έμφαση και προτεραιότητα στην εφαρμογή, στην έμπρακτη εφαρμογή, γιατί έχουμε ήδη πληθώρα οδηγιών και κανονισμών Έχουμε φυστάμενη νομοθεσία. Καλό θα ήταν να δώσουμε έμφαση στην εφαρμογή του, στην πράξη υπάρχει ένα ολόκληρο φάσμα οδηγιών που μένουν ανεφάρμοστε στα κράτη-μέλη. Αν λοιπόν έχουμε επιτέλους μια προεδρία που θα τολμήσει με ουδέτερο τρόπο, χωρίς ε, υπερβολική έγκλη και χωρίς χιλιδί να δώσει έμφαση στην έμπρακτη εφαρμογή των οδηγιών και στην ε, ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, αυτό θα ήταν πραγματικά ευχάριστο. Η κυρία Τζαβέλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σα καλωσορίζω και εύχομαι καλή επιτυχία στην Κυπριακή Προεδρία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ και μερικά χρόνια στην ανατολική πλευρά της Μεσογείου έχουν βρεθεί μεγάλα κοιτάσματα αερίου. Αναφέρουμε κύριε Υπουργέ στο θέμα ε, ε, ασφάλεια εφοδιασμού της, ε, εφοδιασμού της ενεργειακής αγοράς σε ενωσιακό επίπεδο. Έχουν βρεθεί λοιπόν αυτά τα κοιτάσματα. Ήδη το Ισραήλ έχει προχωρεί σε αυτονομία στον ενεργειακό εφοδιασμό και προχωρεί και η, Κύπρο, η Κύπρος εξίσου στην αυτονομία της στον ενεργειακό εφοδιασμό. Το θεωρώ πάρα πολύ πρωτοποριακό αυτό, γιατί ίσως είστε από τα λίγα κράτη-μέλη τα οποία πράγματι μπορούν να αυτοεφοδιάζονται με ενέργεια. Το δεύτερο σημείο είναι ότι η Κύπρος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει εξαιρετικές σχέσεις με όλο τον αραβικό κόσμο και με το Ισραήλ. Αυτό που είπατε για το συνέδριο που θα κάνετε με τους Υπουργούς Ενέργειας ε, της ε, Νοτιοανατολικής ε, Μεσογείου το θεωρώ εξαιρετικό και θα μπορούσε να συμβάλλει ή μάλλον θα συμβάλλει αποφασιστικά με, τα με τις νέες κυβερνήσεις μετά την Αραβική Άνοιξη για να μπορεί να έχει μία προσέγγιση με αυτές η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ερώτημά μου είναι το εξής. <clears throat> Θα προχωρήσετε μέσα σε αυτό το πλαίσιο συνεργασία με αραβικό κόσμο, εφοδιασμός της ευρωπαϊκής ενέργειας, νέες πηγές εφοδιασμού. Θα προχωρήσετε και στην έναρξη του καθορισμού των ΑΟΣ σε αυτή την περιοχή. Δεν είναι μόνο το νότιο κομμάτι της Ευρώπης πρέπει να ξεκαθαρίσει τις ΑΟΣ, είναι και η Αρκτική. Αλλά έχετε την ευχαίρεια να κάνετε μια πρωτοποριακή ενέργεια στο νότο, ούτω ώστε και η Αρκτική να δει πώς πηγαίνετε. Η ερώτησή μου είναι, θα προχωρήσετε σε αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον εφαδιασμό της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Καλωσορίζω και εγώ τον Υπουργό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εγώ σαν Κύπριος Ευρωβουλευτής έχω παρακολουθήσει πάρα πολλές παρουσιάσεις Κυπρίων Υπουργών και αντικειμενικά μιλώντας θεωρώ ότι σε αυτά τα πολύ πρώιμα στάδια η πατρίδα μου αποδεικνύει ότι μπορεί να έχει μια πάρα πολύ επικοδομητική ε, προεδρία όχι μόνο εκ του γεγονότος ότι είναι μικρό κράτος και συνακόλουθα έχει λιγότερες, ε, λιγότερα εθνικά συμφέροντα. Ε, θέλω να υπογραμμίσω αυτό που είπε ο υπουργό ότι επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση προσανατολίζεται όχι μόνο προς την κατεύθυνση της λιτότητας αλλά της ανάπτυξης πια αν και αυτό δεν είναι έτσι πάρα πολύ εμφανές, καθαρό δεν είναι πολύ κρυστάλλινο ε, θέλουμε ακόμα πολλά βήματα για να το δούμε να πραγματοποιείται προς αυτή την κατεύθυνση όμως θέλω να βάλω μία ερώτηση ε, έγινε ευρία αναφορά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπάρχει ένας προτινόμενος προϋπολογισμός 2,5 δισεκατομμυρίων για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να αποτελούν και μερικά εκατομμύρια σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θεωρώ ότι αυτό το ποσό δεν μπορεί να συνδεθεί εύκολα με την έννοια της ανάπτυξης. Ε, υπάρχει τρόπος κατά την άποψη του Υπουργείου σας, της Προεδρίας σας, να αυξηθεί αυτό το ποσό. Ευχαριστώ. Grazie, collega Weber. Και εγώ χαίρομαι για την παρουσία του κύριου Υπουργού. Χαίρομαι και για αυτά που μας είπατε για την αναγκαιότητα να στηρίξουμε, να ευνοήσουμε την επιχειρηματικότητα και τους επιχειρηματίες. Να προωθήσουμε μια νέα γενιά που αναδεικνύεται αυτή τη στιγμή ηγετικών στελεχών επιχειρήσεων στην Ήπειρό μας. Η σημασία που αποδίδεται στην στήριξη και υπεράσπιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι ουσιώδη και για μένα. Αναφερθήκατε στην πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις, Small Business Act, που εγκρίθηκε πριν από τέσσερα χρόνια από την Ένωση. Αλλά δεν βλέπουμε και πολλά πράγματα συγκεκριμένης εφαρμογής. Δεσμευθήκατε να προωθήσετε το θέμα αυτό. Οπότε να θέσω δύο ερωτήσεις για μία από τις πλευρές. Γιατί ε, η πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις θέλει να δίδονται, όπως και στις ΗΠΑ, ένα τμήμα των δημοσίων ε, προμηθειών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αλλά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν μόνο ένα πρόβλημα πρόσβαση στην αγορά. Έχουν και δύο πολύ συγκεκριμένα προβλήματα στην περίοδο κρίσης που ζούμε. Η πρώτη δυσχέρεια είναι η δυσχέρεια χρηματοδότησης το τραπεζικό σύστημα διστάζει ιδιαίτερα να χρηματοδοτήσει γενικά τις επιχειρήσεις και τις μικρομεσές πολύ περισσότερο λόγω του κινδύνου που κάτι τέτοιο θα σήμαινε. Θα έπρεπε λοιπόν να επινοήσουμε ένα συγκεκριμένο, πιο στοχοπροσιλωμένο σύστημα χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το δεύτερο πρόβλημα που έχουν είναι ότι όλο και περισσότερο και με πολύ έντονο τρόπο αντιμετωπίζουν αθέμητο ανταγωνισμό συγκεκριμένα τις απομιμήσεις, κλοπή πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, αλλά και άλλες μορφές του ανταγωνισμού. Και δεν έχουν, αντίθετα με τις ε, μεγάλες επιχειρήσεις, τη δυνατότητα να προσφύγουν σε διαδικασίες προστασίας του ΠΟΕ, γιατί είναι βαριές, κρατάνε πολύ χρόνο και είναι ακριβές μπορούν να απευθυνθούν στον ε, οργανισμό ε, επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ, οι μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά οι μικρομεσαίες όχι. Τι λοιπόν σκοπεύετε να κάνετε για να διευκολύνετε, να βοηθήσετε τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις να προσφεύγουν σε κάποια μορφή νομικής στήριξης κατά των μορφών dumping που υφίστανται. Σας ευχαριστώ η κυρία Μαζέη Κουκόβιτς. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμε κύριε Υπουργέ. Κύριε Σιλικιώτη. Ελπίζω να προφέρω σωστά το όνομά σας. Σας ευχαριστώ σας ευχαριστούμε θερμά για την ε, παρουσίαση, την παρουσία σας και την παρουσίασή σας ε, εδώ. Και θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή επιτυχία, καλή τύχη. Μπορεί να είστε μικρή χώρα, αλλά ευελπιστώ ότι η Προεδρία σας θα είναι καταπληκτική. Είχα και εγώ παρόμοιες εμπειρίες στον τομέα αυτό, όταν η Σλοβενία ανέλαβε το 2008 την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φαίνεται ότι κι εσείς είστε πολύ φιλόδοξη Προεδρία, αλλά δεν βλέπω κάπως πιο συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους πιο απτούς στόχους που να γίνονται πιο εύκολα κατανοητοί και εύληπτοι για τους απλούς πολίτες. Είστε και υπουργό τουρισμού στη χώρα σας. Ποια είναι λοιπόν η γνώμη σας ε, για την ανάπτυξη. Ο τουρισμός είναι πολύ σημαντικός κλάδος και για την ανάπτυξη στην Ευρώπη, για πολλές χώρες όπως ε, τη δική σας. Και νομίζω ότι πολλές χώρες έχουν πολλά να κάνουν στον κλάδο του τουρισμού. Τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε λοιπόν τον τουρισμό για να συμβάλλει περισσότερο στην ανάπτυξη και πώς να διασυνδέσουμε τον τουρισμό με την υγεία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Θα προβλέψετε κάποιες συγκεκριμένες δραστηριότητες για τα διασυνοριακά θέματα υγείας σε μια πρώτη φάση αυτό μπορούσε να οδηγήσει και σε επίδραση στον τουρισμό. Η κυρία Τζόρνταν. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Έχω μερικές σύντομες ερωτήσεις. Πρώτον, ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Είπατε ότι είστε υπέρ του βελτίωσης κατά 20%. Έχουμε μια συμφωνία για 17%. 17% της ενεργειακής αποδοτικότητας στη νέα οδηγία. Συγκεκριμένα λοιπόν προβλέπετε μέτρα για τον τομέα αυτό. Δεύτερον, τονίσατε την ανάγκη μείωσης των εκπομπών και την ε, ενεργειακή ασφάλεια. Είπατε πως είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει σταθερό κλίμα για τους επενδυτές. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να καταλήξουν σε θέση για τον οδικό χάρτη για την ενέργεια το 2050. Είπατε ότι οι νέες πολιτικές πρέπει να σχεδιαστούν με στόχο να συμβαδίζουν με τους στόχους του 2050. Τι σημαίνει αυτό συγκεκριμένα. Θα ήσασταν υπέρ δηλαδή να υπάρξουν νέοι στόχοι. Ποιοι θα ήσαν αυτοί οι στόχοι και θα είναι δεσμευτικοί και κάτι ακόμη. Θα ήθελα να ακούσω την προσωπική σας αντίληψη για το εξής. Στον ε, ενεργειακό οδικό χάρτη αναφέρεται ότι θα υπάρξει διεθνής δράση για την κλιματική αλλαγή. Τι είδους διεθνής δράση. Γιατί δεν ξέρουμε τι θα συμβεί στα διεθνή φόρα. Η Ευρώπη είναι σε κατάσταση κρίσης και πιστεύω ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής μόνοι μας. Και κάτι άλλο. Στόχος μας είναι να υπάρξει μια πλήρως λειτουργική εσωτερική αγορά ενέργειας μέχρι το 2014. Ο οργανισμός ACER θα παίξει ρόλο κλειδί γι' αυτό, αλλά μας είπαν ότι έχουν προβλήματα προϋπολογισμού. Ερώτηση λοιπόν θα τους βοηθήσετε να επιτύχουν τους στόχους τους. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι σε δέκα ερωτήσεις είναι δύσκολο να λάβει κανείς δέκα απαντήσεις γιατί υπολείπονται πέντε λεπτά μέχρι τη λήξη της συνάντησης. Κορέια Ντακάμπος. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ και εγώ τον Υπουργό κύριο Σιλικιώτη, να τον ευχαριστήσω θερμά που ήρθε στην συνεδρίασή μας και κυρίως να το συγχαρώ για το σύνθημα της Κυπριακής Προεδρίας, μια καλύτερη Ευρώπη για τους πολίτες της. Αυτό μας εντυπωσιάζει και μας ικανοποιεί. Επίσης θα ήθελα να εκφράσω την ευαρέσκειά μου για την προτεραιότητα που αποδίδει η Κυπριακή Προεδρία στην άμεση έγκριση του κανονισμού για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας. Εγώ είμαι εισηγητή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό και χαίρομαι για τη φιλοδοξία σας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερος και υπολογίζουμε και περιμένουμε πολλά από την η Προεδρία προκειμένου να προωθήσει την όσο το δυνατόν πιο γρήγορη έγκριση. Στις 28 και 29 Ιουνίου αναφέρθηκε ρητά στο Συμβούλιο αυτό το θέμα, αλλά κρίμα πραγματικά που αναβλήθηκε η έγκριση από την Επιτροπή μας της έκθεσης. Έγινε αναβολή για τη συνεδρία στις 18 Σεπτεμβρίου. Εγώ έμεινα ιδιαίτερα απογοητευμένος αυτή την αναβολή, αλλά ελπίζω το Σεπτέμβριο να το δεκπεραιώσουμε. Θα ήθελα επίσης να σας υπενθυμίσω ότι συμφωνούμε με την διακυβερνητική συνδιάσκεψη για την ενέργεια στην Ανατολική Μεσόγειο, που ελπίζω να ε, αναπτύξετε τις ε, προσπάθειές σας για την ε, εξόρυξη φυσικού αερίου, αλλά υπάρχει έχουμε πρόβλημα ε, γιατί υφιστάμεθα ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον αθέμητο ανταγωνισμό από χώρε που κάνουν ενεργειακό dumping. Ε, και με πολύ μεγάλη ικανοποίηση θα δεχτώ την πρόσκλησή σα στην στο άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο της 17 η Σεπτεμβρίου για τι ανανεώσιμε πηγές ενέργειας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σας καλωσορίζω και εγώ κύριε Υπουργέ. Θα υποβάλω μία ερώτηση σε σχέση με τον τουρισμό. Ξέρετε ότι στο πρόγραμμα COSME ο τουρισμός είναι ένα από τα βασικά προγράμματα που ανακύπτουν, ποιο θα είναι το αποτύπωμα και η πρωτοβουλία που θα αναλάβει η Προεδρία σας αυτό το εξάμεινο. Νομίζω ότι θα μπορούσατε να οριοθετήσετε το θέμα έτσι ώστε ο τουρισμός να αποτελέσει στοιχείο ανταγωνιστικότητας. Ευχαριστώ. Θα είμαι επιγραμματικός. Δεν θα θέσω ερωτήσεις. Κύριε Υπουργέ, θα σας πω ποιες είναι οι δικές μας ανάγκες, ανάγκες ομάδες μας. Ή μιλήσατε για την επιχειρηματικότητα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πολιτική, βιομηχανική πολιτική, αλλά δυστυχώς όλοι αυτοί οι κλάδοι προσβλέπουν σε άμεσο κέρδος και δεν τους ενδιαφέρουν ε, οι ανάγκε του πληθυσμού. Σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίε επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα. Μα οι μικρομεσαίε επιχειρήσεις υπονομεύονται και ε, υποφέρουν κυρίως από την υπερβολική γραφειοκρατία και το χαρτομάνι. Αν δεν δημιουργηθούν ε, νέες διατάξεις για την, ωρα... για την καλύτερη διαφάνεια, για νέους κανόνες με τις τράπεζες, ε, και για την απροθυμία των τραπεζών να βοηθήσουν τι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν πρόκειται να αναπτυχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Θα συνεχίσουν να ε, ταλανίζονται στο μέτρο που δεν υπάρχει δυνατότητα πωλήσεων, γιατί οι πολίτε δεν έχουν αγοραστική δύναμη πια. Σε ό,τι αφορά τη βιομηχανική πολιτική. Πιστεύουμε ότι μόνο η αγορά θα πρέπει να αποφασίσει, ε, ότι η αγορά αποφασίζει ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει. Δεν είναι σωστή αυτή δεν είναι σωστή αυτή η τακτική, δεν θα μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τι ανάγκε των 500 εκατομμυρίων πολιτών. Σε ό,τι αφορά τι ενεργειακέ ανάγκε, λίγη ηθική επιτέλου και λίγη διοντολογία. Δεν μπορούμε να αποθηκεύουμε ηλεκτρική ενέργεια. Όταν τη μεταφέρουμε, έχουμε απώλειε στη μεταφορά. Όμω στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε πολύ μεγαλύτερε πωλήσει ηλεκτρική ενέργεια από ό,τι παραγωγή τη. Φανταστείτε τι κρύβεται πίσω από αυτό. Νομίζω ότι θα πρέπει να απαγορεύσουμε επιτέλους μια τέτοια πολιτική. Ευχαριστώ. Η κυρία Τόγια, τελευταία ομιλήτρια, εντάχει σας παρακαλώ. Καλημέρα σας κύριε Υπουργέ. Εξ ονόματος και της κυρίας Παπαδοπούλου Αντιγόνης λαμβάνω το λόγο γιατί δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να παρέμβει. Ε, οι Κύπροι συνάδελφοι μας ε, εξωθούν προς αυτή, αυτού του τύπου την εργασία. Ως προς το Άτσερ θα ακούσουμε τι έχουν να μας πούν οι ρυθμιστικές αρχές. Έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη σε αυτό το μεγάλο οργανισμό, τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών, Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας και ως προς το κόσμο δέχομαι αυτά που είπε η συνάδελφος για το μέσον αυτό, για την πρόθεση του τουρισμού. Πιστεύετε και εσείς στην εξέλιξη του κόσμου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους Δυστυχώς θα πρέπει να είμαι πιο αυστηρή στο μέλλον. Δεν θα πρέπει να παραβαίνουμε το χρόνο ομιλίας, γιατί διαφορετικά θα βρισκόμαστε σε τέτοια αδιέξοδα. Θα ήθελα να ζητήσω από τον Υπουργό, γνωρίζω ότι δεν μπορεί να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα, και οι συνάδελφοι το κατανοούν πολύ καλά μπορείτε να προσπαθήσετε τουλάχιστον να επικεντρωθείτε στα ε, βασικότερα θέματα κατά τα επόμενα πέντε λεπτά, χωρίς να απαντήσετε μεμονωμένα στους συναδέλφους. Διαφορετικά είναι αδύνατον να απαντήσετε μέσα σε πέντε λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, θα προσπαθήσω έτσι πολύ σύντομα. Βεβαίω υπάρχουν ερωτήματα να ξεκινήσω με το ερώτημα του κύριου Καρβάτσο για την πυρηνική ενέργεια. Είναι το γεγονό ότι οι επιπτώσει από τα πυρηνικά συμβάντα συχνά δεν έχουν τοπικού ούτε χρονικού περιορισμού, ξεπερνούν από οποιαδήποτε σύνορα. Χρειάζεται και στην Ευρώπη να αλλά και με του γείτονε μα να υπάρχει συνεργασία. Είναι σημαντικό το ότι αυτή τη στιγμή προωθείται το stress test σε 140 πυρηνικού σταθμού. Είναι κάτι που συνεννόμαστε με την Επιτροπή και θα δούμε τα αποτελέσματα για να δούμε και τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να πάρουμε και βεβαίως παράλληλα ε, δίνουμε σημασία στο πώς θα αναπτύξουμε ε, εναλλακτικέ μορφές ενέργειας ε, όπως είναι ανανεώσιμες πηγές, όπως είναι βεβαίως η αξιοποίηση του φυσικού αερίου που είναι καθαρότερη μορφή ενέργειας. Για τα θέματα της ανταγωνιστικότητας να πω ότι και των επιχειρήσεων να πω ναι πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έφαση, ε, μερικοί ε, ευρωβουλευτέ έβαλαν αυτό το θέμα, πρώτα-πρώτα τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για το πρόγραμμα COSME, ένα ζήτημα αυτό που χρειαζόμαστε είναι επιχειρήματα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μέρο του πολιετέ δημοσιονομικού πλαισίου, όπω είπε και η κυρία Βαν Πρόεμπτ, και ε, χρειάζεται εδώ να έχουμε επιχειρήματα για να δούμε πώ θα καταφέρουμε μέσα σε αυτόν τον καταμερισμό, μέσα σε αυτή τη συζήτηση, ενδεχομένω να υπάρχει ε, μεγαλύτερη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Συμφωνώ αυτά που έθεσαν μερικοί ευρωβουλευτέ για τα θέματα γραφειοκρατία. Βεβαίω, ένα θέμα που συζήτησα χθε στην Επιτροπή ΙΚΟ είναι τα ζητήματα των δημόσιων συμβάσεων, πώ περιερίζομαι τι γραφειοκρατικέ ρυθμίσει, πώ διευκολύνουμε την πρόσβαση στι δημόσιε συμβάσει των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι μικρομεσαίε επιχειρήσει είναι η ραχοκαλιά τη οικονομία τη Ευρώπη ε, και χρειάζεται και συγκεκριμένα προγράμματα, αλλά χρειάζονται και μέσα από τις διαδικασίες μας να διευκολύνουμε τη δική τους πρόσβαση. <clears throat> Αυτά που αφορά τον αθέμητο ανταγωνισμό που τέθηκε από κάποιους ευρωβουλευτές, βέβαια είναι αυτά ζητήματα που αφορούν τις εμπορικές συμφωνίες. Είμαι και υπουργό ε, ε, αρμόδιος για αυτά τα θέματα. Το απόγευμα θα είμαι στην Επιτροπή ΝΙΤΑ, όπου θα συζητήσω βέβαια το πρόγραμμα του επόμενου εξαμένου. Χρειάζεται ε, να υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες σε αυτές τις εμπορικές συμφωνίες, ώστε να μην έχουμε αυτά τα φαινόμενα που αναφέρθηκαν μερικοί <clears throat> ευρωβουλευτές. Ε, τώρα, στα ζητήματα ε, για τα προγράμματα και το πόσο <clears throat> φιλόδοξοι είμαστε, η κυρία Ρώτη έθεσε βέβαιο στο θέμα ότι η έμπρακτη εφαρμογή και τέθηκε και από, τον, και από άλλον Ευρωβουλευτή, νομίζω ότι εκείνο που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι η συνεργασία όλων μας για να μπορέσουμε να πρώτα-πρώτα να προωθήσουμε πιο γρήγορα συγκεκριμένες οδηγίες. Δηλαδή η οδηγία <clears throat> για τις ε, ενεργειακές υποδομές είναι σημαντική γιατί δεν διασφαλίζει μόνο ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Δίνει δυνατότητα να προχωρήσουμε στην υλοποίηση αναπτυξιακών έργων που θα δώσουν όθηση και στην ανάπτυξη, αλλά θα δημιουργήσουν ε, και θέσει εργασία. Παράλληλα, χρειάζονται βεβαίω καλύτεροι μηχανισμοί <clears throat> για υλοποίηση όλων αυτών που <clears throat> εγκρίνομαι. Ε, στα θέματα που έθεσε ο, ο κύριος Βέμπερ νομίζω έχω απαντήσει για τις δημόσιες προμήθειες. Ε, έρχομαι τώρα σε κάποια ζητήματα επιμέρους. Οι στόχοι καταλαβαίνουν καμιά φορά ότι ε, για να πάμε στον οδικό χάρτη να υλοποιήσουμε του στόχου που θέτουμε το 2050, πρέπει να θέσουμε διάμεσου στόχου. Και αυτό είναι η αναφορά ότι θα πρέπει να θέσουμε και στόχου για το 2030. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο. Ναι, κατανοούμε τι δυσκολίε που υπάρχουν σε πολλά κράτη-μέλη και αναφέρομαι στι οικονομικέ δυσκολίε. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ευέλικτοι στην εφαρμογή ε, αυτών των στόχων. Όμω, δεν μπορούμε από το να έχουμε στόχους και να επιδιώκουμε τους στόχους. Έτσι θα βοηθήσει ε, να ε, εισαγάγουμε και ε, περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρισμού και στη μείωση των εκπομπών αερίου και στην καλύτερη ενεργειακή απόδοση. Ε, <clears throat> ήθελα να θέσω και τα ζητήματα, ακόμα δύο ζητήματα που θέθηκαν. το ένα αφορά Βέβαια, στο ε, τι γίνεται στην Ανατολική Μεσόγειο, αντιλαμβάνεστε ω ε, Κύπρο Υπουργό, είναι ε, στη δική μας τη χώρα που, ε, κοντά που γίνονται αυτές τι εξελίξεις, Θα ήθελα να σημειώσω δύο πράγματα μόνο. Χρειαζόμαστε να ενισχύσουμε την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Στην Ανατολική Μεσόγειο, με τι νέε ανακαλύψεις που υπάρχουν, υπάρχει δυνατότητα να δημιουργήσουμε έναν τρίτο διάδρομο ενεργειακής τροφοδοσίας τη Ευρώπη σε συνεργασία βεβαίω με τι χώρε τη περιοχή. Και αυτό είναι θετικό γιατί <clears throat> η Κύπρος είναι κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορεί να είναι έξω από τι προτεραιότητε τη η ανάγκη να ενισχύσει στο μέτρο των δυνάμεων του βέβαια την ενεργειακή ασφάλεια τη Ευρώπη ε, και βεβαίω να διευρύνουμε τη συνεργασία. Είναι θετικό το γεγονό αυτό που αναφέρθηκε και η κυρία Τσαβέλλα ότι η Κύπρος έχει άρεστε σχέσει με του γείτονε τη και αναφέρομαστε και στο Ισραήλ και στου Άραβε γειτονέ μα. Παράλληλα, είναι σημαντικό μαζί με του γείτονε μα και στην Ανατολική Μεσόγειο και στι άλλε περιοχέ τη Μεσογείου και στη Βόρεια Θάλασσα να δούμε τρόπου συνεργασία για να υπάρχει ασφάλεια στι ε, γεωτρήσει. Ε, μιλούμε για ιδιαίτερα η Μεσόγειο είναι μια κλειστή θάλασσα και αυτού, σε αυτόν τον στόχο ε, προσλέπει η πρωτοβουλία μα να συνεργαστούμε με του γείτονε μα. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση στη συνεργασία με του γείτονε τη πρέπει να δημιουργήσει ε, συμφωνίε, σύμφωνα για να υπάρξει ασφάλεια προστασία τη θάλασσα, προστασία του περιβάλλοντο. Ε, <clears throat> σε ό,τι αφορά τα θέματα του τουρισμού, ε, είναι σημαντικό να πω ότι η Ευρώπη μπορεί και ο στόχος ε, να γίνει ξανά ο ορκιστικότερος προορισμός τουρισμού στον κόσμο. Έχουμε όλα τα δυνατότητα, όλες τις δυνατότητες. Και το περιβάλλον και τις υπηρεσίε ε, και ε, αν θέλετε την ιστορία και την παράδοση. Χρειάζεται εδώ να λειτουργήσουμε περισσότερο ενία. Ένα θέμα που ε, πρέπει να λύσουμε είναι να δούμε, βεβαίω εδώ χρειάζεται να συνεργαστούμε ε, και με την Επιτροπή, είναι η απλοποίηση της διαδικασίας ό,τι αφορά τις θεωρήσεις διαβατηρίου. Υπάρχουν από πολλές νέες αγορές που πρέπει να βρούμε τον τρόπο να διευκολύνουμε δηλαδή την πρόσβασή του στην Ευρώπη. Το δεύτερο είναι οι δυνατότητε για να αναπτύξουμε ε, ε, θεματικό τουρισμό και στην Ευρώπη έχουμε τα χέρια να προσφέρουμε ποιοτικό θεματικό τουρισμό. Είναι κάτι σημαντικό που ανάφερε η κυρία Κούκοβιτ ό,τι αφορά ε, και τον τομέα τη υγεία, και βεβαίω πρέπει να υπάρξει και διασυνοριακή συνεργασία. Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που έθεσε η κυρία Τζόρταν, απλώ επειδή είναι κάπω επιμέρου θέλω να το αναφέρω αυτό, ε, σε ό,τι αφορά την εσωτερική αγορά ενέργεια. Ναι, πρέπει να προωθήσουμε την εσωτερική αγορά. Υπάρχουν ακόμα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι απομονωμένα από τα δίχτυα ενέργεια τη Ευρώπη. Και ε, ακριβώ Πρέπει να υλοποιήσουμε το στόχο μέχρι το 2000 να ολοκληρώσουμε την εσωτερική αγορά μέχρι το 2014 και μέχρι το 2015 να μην υπάρχουν κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, από μονομένα. Και ε, ε, να πω επίσης ότι το θέμα αντιρρυθμιστικών αρχών ενέργειας που έθεσε η κυρία Τόια ε, είναι σημαντικό να ενισχύσουμε τον ρόλο των ανεξάρτητων ρυθμιστικών αρχών ενέργεια, για το ότι κάνουμε δεν φτάνει να έχουμε μηχανισμούς κρατικούς, πρέπει να έχουμε μηχανισμούς ανεξάρτητους, οι οποίοι να λειτουργούν ω σύμβολοι στον τομέα της ενέργειας, αλλά ως αρχές που ρυθμίζουν τα θέματα ενέργειας και ως αρχές που ελέγχουν για να μπορούμε να κάνουμε ε, καλύτερα τη δουλειά μας, ιδιαίτερα στην υλοποίηση των κανονισμών και των οδηγιών της όνωσης, που εδώ πρέπει να είναι ο στόχος όλων μας. Ε, ήθελα να σας ευχαριστήσω για όλες αυτές τα ερωτήσεις και να σας διαβιώσω ότι ε, αυτό που είπε ε, η, η, κυρία Βαν Πρέπτ είναι ότι ναι, η Κύπρος μπορεί να είναι ένας αξιόπιστος διαμεσολαβητής ως ε, μικρή χώρα σε όλα αυτά τα ζητήματα που συζητούμε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Σε ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ. Θα τα ξαναπούμε. Και τώρα θα έχουμε τους δύο επόμενους ομιλητές. Συνεχίζουμε τις εργασίες μας γιατί έχουμε καθυστερήσει κατά 10 λεπτά. Παρακαλώ να φύγουν, να αποχωρήσουν από την αίθουσα όσοι το επιθυμούν. Εντάχει ήθελα να καλωσορίσω τον Λόρδο Μόγκ, τον πρόεδρο του Συμβουλίου Ρυθμιστικών Αρχών και τον Αλμπέρτο Ποτότσνιχ, διευθυντή, που θα μας παρουσιάσουν το σχέδιο προγράμματος εργασίας του οργανισμού αυτού του ΆΣΕΡ για το 2013. Στη συνέχεια, μετά από αυτή τη συνάντηση, προβλέπεται μία συνεδρίαση εργασίας που διοργανώνει το ΆΣΕΡ για όποιον θελήσει να συμμετάσχει. Αρχίζουμε με τις εργασίες μας. Θα έχουμε καταρχήν ε, μία παρουσίαση από το Λόρδο Μόγκ του ρυθμιστικού αυτού φορέα. Έχετε το λόγο. Madam Chair. Πρόεδρε, κύριε και κύριοι, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ γιατί μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω ενώπιον σας. Ξέρω ότι πρέπει να είμαι σύντομος και θα το πράξω πριν δώσω το λόγο στο Διευθυντή. Καταρχήν, η, ως προς το βαθμό συνεργασίας, επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και τον φορέα μας που είναι κρίσιμη σημασίας για το μέλλον, για τις ε, διευθετήσεις του τομέα ενέργειας. Εγώ είμαι επικεφαλής του Διοικητικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Ρυθμιστών. Έχουμε 150 εθνικές, εθνικούς ρυθμιστές που συμμετέχουν στον ευρωπαϊκό αυτό οργανισμό μέσα στα πλαίσια της νομοθέτησης και μας βοηθούν και έμπρακτα και σε πρακτικά ζητήματα. Υπάρχει συμπληρωματικός χαρακτήρας ε, στην εργασία αυτή, δηλαδή από πλευράς Acer του ρυθμιστικού αυτού φορέα αυτού, συντονισμού των ρυθμιστικών αρχών και του Συμβουλίου. Και ένα από τα θέματα που μας απασχολούν είναι η πολιτική υπέρ των καταναλωτών. Το μέλλον διαγράφεται θετικό, αλλά παράλληλα ελοχεύουν και κίνδυνοι. Ο δόκτωρ Τζόρνταν μίλησε για ένα θέμα πόρων και χρηματοδότησης και ο Διευθυντής θα σας μιλήσει για τις επερχόμενες εργασίες. Ελπίζουμε να περάσουν ορισμένα νομοθετήματα που θα μας βοηθήσουν γιατί είχαμε και πρόσφατες αλλαγές με βάση το ενεργειακό πακέτο και ελπίζω ότι θα μας υποστηρίξετε. Ο διευθυντής μας λοιπόν θα σας ε, μιλήσει για ένα πρόγραμμα προκλήσεων ε, το οποίο ελπίζουμε να είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό για το μέλλον. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο κύριος Ποτότσνικ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα συνεχίσω στα αγγλικά. Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα να πω ότι έχουμε να κάνουμε με ένα πρόγραμμα προκλήσεων το οποίο αφορά τον ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο του οργανισμού αυτού η οποία ήταν αναπόσπαστο μέρος του τρίτου πακέτου. Έκτοτε όμως έχουμε επιπρόσθετες ευθύνες και καθήκοντα μέσα στα πλαίσια του REMIT, δηλαδή του κανονισμού για την ακαιρεότητα και διαφάνεια στην ενεργειακή αγορά, το οποίο τώρα συζητείται στο Κοινοβούλιο και ε, από την Ευρωπαϊκή Επίτροπη με βάση επιπρόσθετα καθήκοντα μέχρι το τέλος του 2012. Ε, άρα επεκτείνεται ο, ο ρόλος της όπως ανέφερε και ο Λόρδος Μοκ. Ας δούμε τις προτεραιότητες για το επόμενο έτος, για το 2013 θα μιλήσω λεπτομεριακά και για τις μεμονωμένες δραστηριότητες, αλλά για να οριοθετήσω το όλο ζήτημα, θεωρούμε ότι υπάρχουν θέματα ε, ύψης της σημασίας. Θέλουμε να συμπληρώσουμε την εργασία των κατευθυντηρίων γραμμών πλαισίωσης πριν μπούμε σε επιμέρους προγράμματα. Πρόκειται για κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες έχουν εγκριθεί και αποτελούν το νομοθετικό πλαίσιο μέσα στα πλαίσια του οποίου μπορεί να λειτουργήσει η αγορά ενέργειας μέχρι το 2014. Επίσης θα ε, προωθήσουμε και τον κανονισμό για την ακαιρεότητα και τη διαφάνεια με βάση τα ε, κριτήρια που διαγράφονται. Και θα επανέλθω στο REMIT, στον κανονισμό αυτό. Θέλουμε να επεκτείνουμε τις δραστηριότητες εποπτείας που ξεκίνησαν φέτος με την ε, πρώτη δημοσίευση των περιφερειακών πρωτοβουλειών και θα θέλαμε η ενεργειακή αγορά πραγματικά να καταστεί λειτουργική. Θα πρέπει να θέσουμε σε εφαρμογή και τον κανονισμό REMIT για την ακαιρότητα και τη διαφάνεια και τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για το TEN-E μέσα στα πλαίσια των προγραμμάτων κοινοτικού ενδιαφέροντος. Το πρόγραμμα αυτό είναι διαθέσιμο και, στο, ε, και στην ιστοσελίδα μας και έχετε όλες τις λεπτομέρειες για του χρόνου προβλέπουμε νέες δραστηριότητες, νέους δηλαδή ε, κωδικούς δικτύου, οι οποίοι θα τεθούν σε εφαρμογή ήδη από το 2012. Μέχρι του χρόνου όμως θα έχουμε 12 δίκτυα, τα οποία θα ισχύσουν μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας επιτροπολογίας. Δεν θα ήθελα να μπούμε σε νέους τομείς ως προς τις κατευθυντήριες γραμμές, αλλά θα μπούμε και σε θέματα τιμολόγησης, γιατί είναι θέματα τα οποία σχετίζονται με το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων μέσα στα πλαίσια και των πρωτοβουλειών που θα οριστούν. Θα λάβουμε το σχέδιο ε, Ω προς το δεκαετέ πρόγραμμα ανάπτυξη δικτύων, φέτος το λάβαμε για τα ε, δίκτυα ηλεκτροδότησης. Επίσης, θα πρέπει να ορίσουμε μία πρόταση μέσα στα πλαίσια του Inter-TSO, δηλαδή ε, των διαχειριστών δικτύου μεταφοράς, και σας μίλησα και για την έκθεση εποπτείας και σε επίπεδο περιφερειακό καθαρά. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα διαχειριστούμε τις εξαιρέσεις και τις πιστοποιήσεις καθώς και τις εξαιρέσεις που προβλέπονται, τις απαλλαγές. Σε σχέση με το REMIT, τον κανονισμό αυτό για την ακαιρότητα και τη διαφάνεια στην ενεργειακή αγορά, Έχουμε κατευθυντήριες γραμμές και θα πρέπει να υπάρχει μία κοινή μεθοδολογία και διαφάνεια για τους συμμετέχοντες στην αγορά, για τους εμπλεκόμενους φορείς. Θα πρέπει να υπάρχει μία μεθοδολογία εποπτείας και να λαμβάνουμε υπόψη και τα διάφορα μέσα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών σε σχέση με τις, τα έργα αυτά υποδομών έχουν αρχίσει παρόλο που συζητείται ακόμα ο κανονισμός και συνεργαζόμαστε και με την Επιτροπή έτσι ώστε να ενισχυθεί ο ρόλος της Acer σε προγράμματα κοινού ενδιαφέροντος όπου θα πρέπει να υπάρχουν συνεκτικά κριτήρια και σε περιφερειακό επίπεδο και σε εξατομικευμένο και υπάρχει και το μεθοδολογικό ε, κριτήριο σε σχέση με το, με την, το σχετισμό κόστους ωφελίας. Αυτές είναι και οι βασικές δραστηριότητες. Τώρα θα ήθελα να δούμε τους κινδύνους και την, όπου υπάρχει ε, ανασφάλεια, έλλειψη ασφάλειας και να δούμε που θα μπορέσουμε να δράσουμε με βάση το χρονοδιάγραμμα που διαθέτουμε. Όπως ε, ανέφερε και ο Λόρδος Μόγκ, λαμβάνουμε υπόψη τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές οι οποίες μας υποστήριξαν και θα εξακολουθήσουν να μας υποστηρίζουν. Πολλές από αυτές βεβαίως έχουν να αντιμετωπίσουν την δημοσιονομική λιτότητα και γι' αυτό ίσως η υποστήριξη να μην είναι η ίδια στο μέλλον από τις εθνικές Εθνιστικές αρχές. Ίσως ε, να υπάρξουν ελλείψεις για το νέο έργο μας και θα πρέπει βεβαίως να προσελκύσουμε και εξειδικευμένο προσωπικό. Ως προς τις ε, προκλήσεις και το νέο έργο μας θα πρέπει να εφαρμόσουμε το REMIT, τον κανονισμό αυτό για τη διαφάνεια στην ενεργειακή αγορά ιδιαίτερα. Δεν υπάρχει πείρα στο REMIT, στον κανονισμό αυτό και προβλέπουμε περισσότερο προσωπικό. Ήδη σας είπα στο παρελθόν ότι θέλαμε 15 επιπρόσθετους υπαλλήλου για την εφαρμογή του REMIT, του κανονισμού αυτού για την ενέργεια. Για το 2012-2013 η Επιτροπή προβλέπει 15 υπαλλήλου για την χρήση του συστήματος, αλλά το θέμα παραμένει ανοιχτό για το κατά πόσο θα μπορέσει να καταστεί λειτουργικό με τόσο περιορισμένο προσωπικό. Επίσης, ε, υπάρχουν περικοπές κατά τρεις υπαλλήλου από τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό του 2013. Από πλευράς προϋπολογισμού για την επόμενη χρήση, το σχέδιο προϋπολογισμού που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει πει μείωση 3 εκατομμύρια σύμφωνα με τις προβλέψεις μας και ε, λαμβάνοντας υπόψη τα συνολικά πόσα θα πρέπει να μειώσουμε το λογισμικό για το REMIT και γι' αυτό νομίζω ότι το REMIT, ο κανονισμός για την ενεργειακή αγορά, θα γνωρίσει καθυστερήσεις. Ως προς τη συνεργασία θα ήθελα να πω ότι βασιζόμαστε στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής ε, συνειδητοποίησαν ότι χρειάζονται επιπρόσθετη πόρη και αυτό είναι πολύ καλό για τον οργανισμό, αλλά το πώς μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, αυτό δεν είναι καθόλου σαφές. Ήδη σας είπα ότι το Συμβούλιο κατά τη γνωμοδότησή του στο σχέδιο του ε, μίλησε για μείωση κατά τρεις υπαλλήλου. Αυτές είναι οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά όπως καταλαβαίνετε η ευελιξία έχει και τα όρια της. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ε, παρουσίαση ε, γνωρίζω ότι έπρεπε να περικόψετε κατά πολύ την παρουσίασή σας. Ας δούμε κατά πόσο έχουμε χρόνο για απαντήσεις, ερωτήσεις και απαντήσεις. Ο κύριος Κορέια Ντοκάμπος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. και τον Λόρδο Μοκ και τον Αλμπέρτο Ποτότσινικ που ήρθε στην Επιτροπή μας. Ε, με ιδιαίτερη ικανοποίηση ακούσαμε τις φιλοδοξίες σας και παρακολουθήσαμε και τα προβλήματά σας. Θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία-τέσσερα θέματα. Φυσικά να γνωρίζουμε το έργο του οργανισμού αυτού. Ε, εγώ χρειάστηκε να εξοικειωθώ με το θέμα αυτό και διαπιστώνω ότι πραγματικά το έργο του οργανισμού είναι τελείως ανεξάρτητο και είναι σημαντικό να έχουμε ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές που θα χαίρουν σεβασμού στην αγορά. Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι χρειαζόμαστε πιο σημαντικά βήματα στο μέλλον και γνωρίζω ότι είμαι εισηγητής ε, και για τα, τους κώδικες των δικτύων και τις ε, κατευθυντήρες γραμμές του πλαισίου θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειές μας και να συμπληρώσουμε τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να εφαρμόσουμε μία μέθοδο για την καλύτερη εκτέλεση και εφαρμογή αυτών των κωδίκων των δικτύων. Και φυσικά προσβλέπουμε στο ε, σημαντικό ρόλο του οργανισμού σας στο μέλλον για, τις, ε, για τα ναύλα μετα, μεταφοράς. Σε ό,τι αφορά τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας και την επιλογή ε, προγραμμάτων κοινού ενδιαφέροντος. Νομίζω ότι είναι τεράστιο αυτό το έργο, τιτάνιο, κολοσιαίο, δεν θα πρέπει να έχουμε ψευδεστήσεις, θα χρειαστούν τεράστιες προσπάθειες, θα γίνουν σφοδρές συζητήσεις, ίσως και κάποιες αντιπαραθέσεις. Σε ό,τι αφορά το TNPDP για το φυσικό αέριο, και ολοκληρώνω κυρία Πρόεδρε, χαίρομαι ότι θέλετε καλές σχέσεις με τους TSOs. Είναι σημαντικό ρυθμιστικές αρχές και TSOs να έχουν αγαστές σχέσεις και επίσης να αναγνωρίσω ότι παρά το δύσκολο έργο σας ε, θα ήθελα να εκφράσω την ε, ε, συμπάθεια μου και τη συμπαράστασή μου για τα αιτήματά σας <laughs> αλλά πέραν της συμπαράστασης δεν μπορώ να κάνω τίποτα παραπάνω. Ευχαριστώ. Η κυρία Τζόρνταν. Και εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να μειωθεί η απόσταση ανάμεσα στην νομοθεσία που εγκρίνουμε και τι εφαρμόζεται στην πράξη. Νομίζω ότι η εφαρμογή του κανονισμού REMIT είναι θεμελιώδους σημασίας. Δεν θα έχουμε η εσωτερική αγορά σε αυτό το τομέα μέχρι το 2014 εάν δεν γίνει κάτι τέτοιο. Η Επιτροπή απάντησε στην ερώτησή μου, θέλω να σε ενημερώσω. Σύμφωνα με τη νέα πρόταση, 8,8 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν στον οργανισμό σας, τρία εκ των οποίων ε, πρέπει να δοθούν αποκλειστικά στο REMIT. Ε, είναι διαφορετικά τα στοιχεία από αυτά που μας είπατε την τελευταία φορά που ήσασταν στην Ήτρε, γι' αυτό θα ήθελα τα σχόλιά σας. Από το Συμβούλιο όμως δυστυχώς δεν έχω πάρει ακόμα επάντηση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τούρμας. Θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε σήμερα αλλά και αύριο είναι επανεξέταση της εσωτερικής αγοράς. Υπάρχει μια μεταρρύθμιση της ε, αγοράς ηλεκτρισμού στις ΗΠΑ, στη Γαλλία επίσης, αμφίβολες καταστάσεις. Άρα θα υπάρξουν προβλήματα όσον αφορά τις εθνικές αγορές και τη χωρητικότητά τους. Πρέπει να καταδείξουμε τα αποτελέσματα μιας ε, ενιαίας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Και για αυτά που είπατε για τον προϋπολογισμό, πρέπει να δείξουμε στα κράτη-μέλη ότι όσο πιο ενοποιημένη είναι η εσωτερική αγορά, τόσο περισσότερο κερδίζουν οι καταναλωτές. Με μερικά επιπλέον εκατομμυριάκια για το Acer που θα το καταστήσει δυνατό, θα αποδώσουν τεράστια, πολύ περισσότερα κέρδη. Μήπως θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποια στοιχεία για να τεκμηρώσουμε αυτές τις ε, ε, ε, θέσεις μας. Για το ρήμι τώρα. Ξέρουμε ότι υπάρχει, εγκληματικότητα, υπάρχει το φαινόμενο της εγκληματικότητας των στελεχών επιχειρήσεων. Εάν επιτρέψουμε κάτι τέτοιο, θα χάσουμε την ε, αξιοπιστία μας. Πρέπει λοιπόν να ξαναποδείξουμε ότι το ACEA e χρειάζεται αυτούς τους πόρους και η Επιτροπή μας θα πρέπει να πείσει τους ε, συναδέλφους μας στην Επιτροπή Προϋπολογισμών ότι μερικά μόνο εκατομμύρια για το Acer πρέπει να είναι και για αυτούς προτεραιότητα όταν αρχίσουν να διαπραγματεύονται με τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Μπαντή, ακούσε. Ευχαριστώ για την παρουσία σας, την παρουσία του προγράμματος εργασίας σας να αποφελθώ από την ευκαιρία για να κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση που μας ανησυχεί κάπως, μας απασχολεί κάπως. Θα μάθατε ότι η Ισπανική κυβέρνηση εδώ και μερικούς μήνες ανήγγειλε την πρόθεσή της να υπάρξει μία μόνο επιτροπή όπου θα συνενωθούν όλοι οι οργανισμοί και όλες οι επιτροπές που ασχολούνται με την ε, σωστή λειτουργία της αγοράς σε διάφορους τομείς πολύ ευαίσθητους όπως είναι η τηλεπικοινωνίες και ενέργεια. Και υπάρχει ένα νομοσχέδιο που θέλει να επανεθνικοποιηθούν, να υπάρξει δηλαδή συγκέντρωση των διαφόρων οργανισμών που τώρα λειτουργούν σε περιφερειακό επίπεδο. Θα δημιουργηθεί λοιπόν ένας οργανισμός συντονισμού. Πώς εκτιμάτε εσείς αυτή την Ισπανική πρωτοβουλία να δημιουργηθεί αυτός ο οργανισμός που θα είναι ένας ε, καθολικός ρυθμιστής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη αν... εκφράστηκε από αυτού με κάποια ανησυχία. Ευχαριστώ τελευταίος, ο Σάνθος Πρώτη. Εντάχει και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσίασή σας. Θεωρώ ότι αποτελεί άμεση ανάγκη η ύπαρξη ενός διευρωπαϊκού δικτύου, διότι μόνο με αυτό ραχοκοκαλιά θα μπορέσουμε να βελτιστοποιήσουμε όλες τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες θα πρέπει να είναι και συμβατές. Δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά θα ήθελα το δικό σας σχολιασμό να μου πείτε δηλαδή πώς μπορούμε να φτάσουμε σε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ποτόσμικ. Ευχαριστώ. Να απαντήσω μερικέ και μετά ο Λόρδος Μόγκ θα συνεχίσει. Στον κύριο Ντεκάμπος συμφωνώ ότι του χρόνου θα αντιμετωπίσουμε μια ιδιαίτερα σημαντική πρόκληση. Προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε τους κώδικες δικτύων που θα είναι η νομική βάση για την ε, ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, της εσωτερικής αγοράς. Αλλά έχουμε και τις νέες καθεντήρες γραμμές για την διευρωπαϊκή υποδομή ενέργειας. Μεγάλη πρόκληση λοιπόν για τον οργανισμό μας. Είναι νέο να αντιμετωπίσει ευνοϊκά το θέμα μου. Ο Λόρδος Μόγκ. Με συγχωρείτε. Σε αυτό που είπε ο κύριος Τούρμες, ήμουν υπεύθυνο για την ε, ανάπτυξη της ενίας αγοράς όταν ήμουν στην Επιτροπή. Άρα μπορώ να δω και τα ωφέλη αλλά και τις εντάσεις που προκύπτουν στην προσπάθεια επίτευξης αυτού του στόχου. Βεβαίως, οπωσδήποτε, πρέπει να υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα ότι θα έχουμε ωφέλη από την ε, ενιοποίηση της αγοράς. Διότι οι χώρες που θα συνεργάζονται θα ελαχιστοποιούν ε, το ενδεχόμενο επεισοδίων και διακοπών Προς το παρόν έχουμε επαρκή ενέργεια, αλλά στο μέλλον μπορεί να υπάρχουν ελλείψεις. Αλλά ε, να προειδοποιήσω κιόλα. Εάν σας δημιουργήσουν την εντύπωση ότι η κατάσταση ε, ε, δεν προχωράει αυτή τη στιγμή, ότι υπάρχει στασιμότητα, δεν είναι σωστή εντύπωση. Ε, υπάρχει πορεία προς τα μπρος, υπάρχει πρόοδος, χρειαζόμαστε περισσότερους πόρους, αλλά δεν είναι η συνολική εικόνα αυτή. Και βεβαίως ε, είμαι απόλυτα πεισμένος ότι χρειάζεται ενιαία αγορά και στην ενέργεια. Δεν θα σχολιάσω τα σχόλιά σας για την ε, κατάσταση στον στο Βασίλειο. Για την κυρία Μπάτια. Βεβαίως οι ρυθμιστές δεν είναι σε θέση να σχολιάζουν την κατάσταση σε ένα κάποιο κράτος μέλος, γιατί αυτό είναι ευθύνη της κυβέρνησης του κράτους αυτού και η Επιτροπή, αν θέλει να προσφύγει κατά κάποιου κράτους μέλους, είναι σε θέση να το κάνει. Αλλά τονίζω ότι έχουμε αρκετά στοιχεία, ότι υπάρχει περισσότερη συνεργασία και περισσότερη κατοχήρωση της λειτουργίας διάφορων ρυθμιστικών αρχών. Η ανησυχία είναι πρώτα απ' όλα να υπάρχει ανεξαρτησία, δεύτερον αρκετή εθνική πόροι για τους εθνικούς ρυθμιστές και τρίτον να υπάρχει δυνατότητα χορήγηση, ε, μάλλον οι κυβέρνησεις να έχουν δυνατότητα να παρέχουν ε, συμβουλές σε αυτές τις ε, ρυθμιστικές αρχές και αντιστρόφως, αλλά να μην υπάρχει έλεγχο. Είμαι σίγουρος ότι η Επιτροπή θα κάνει ό,τι μπορεί, ούτω ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα στην Ισπανία του ερχόμενου μήνε. Και από πλευρά του κ. Ποτόσνη και μου του ιδίου ευχαριστώ την Επιτροπή σα για το χρόνο σα. Ξέρω ότι είχατε πολλά θέματα. Ελπίζω να μην σα απασχολήσαμε υπερβολικά. Σα ευχαριστώ για την παρελθούσα και, προβλέπω και προσβλέπω και στην μελλοντική υποστήριξή σα. Ευχαριστούμε πολύ τον Πρόεδρο και τον Διευθυντή του Συμβουλίου Ρυθμιστικών Αρχών για τη διαθεσιμότητά τους για την παρουσία τους. Ε, ευχαριστεί η Πρόεδρος τους Διερμηνείς. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση της Επιτροπής της 3 το απόγευμα. Γεια σας.